Good morning. Καλημέρα σας. Σας συνεχίσω στα πορτογαλικά. Bon dia a ε, todos. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να καλημερίσω και τους συναδέλφους που έρχονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια και τους συναδέλφους από την Επιτροπή Νομικών ε, Θεμάτων και από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών. Πρόκειται για μια κοινή συνεδρίαση αυτών των δύο επιτροπών. Το πρώτο σημείο της ημερήσία διάταξης είναι η έγκριση της ημερησία διάταξης αν ε, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρώ ότι εγκρίνεται. Τώρα, σημείο 2. Ανακοίνωση, ανακοινώσεις του Προέδρου ή της Προέδρου. Δεν ε, έχω εγώ κάποια ανακοίνωση να κάνω εδώ. Και να περάσουμε στο σημείο 3. που είναι η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την έκθεση της κυρίας Εβελίν Ρέγνερ και της κυρίας Ρόβι Κράτσα για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φίλων σε θέσεις με εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εταιριών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Peço Λοιπόν, πριν ah, να δώσω το λόγο στην εισηγητρία, η κυρία Ρέγκνερ θα πάρει το λόγο ως ε, πρόεδρος ε, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. das ganz einfach. Unkompliziert. So. Nein, nein, das geht schon. Oh, voilà. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt... Κυρίες και κύριοι, τώρα δουλεύουν τα μικρόφωνα, από ό,τι φαίνεται. Θα ήθελα εκ μέρους της Επιτροπής των Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από πλευράς μου να σας καλωσορίσω και εγώ. Έχουμε μια ακρόαση σήμερα η οποία αφορά και τις δύο επιτροπές μας, την Επιτροπή των Γυναικών και την Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων και αφορά σημαντικά και για τις δύο επιτροπές ζητήματα. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φίλων των ανδρών και γυναικών, δηλαδή σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. Πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τις συζητήσεις μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αλλά βεβαίως και πάνω απ' όλα πάρα πολύ σημαντικό και για τις συζητήσεις που αναπτύσσονται στα κράτη-μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια. Και γι' αυτό εδώ έχουμε οργανώσει την κοινή ε, συνεδρία των δύο επιτροπών με την εκπόνηση κοινή εκθέσεως και θέλουμε να ακούσουμε σήμερα τη δική σας γνώμη, τις δικές σας γνώμες και να συζητήσουμε το θέμα αυτό μαζί σας. Εν συντομία, θα ήθελα να παρουσιάσω το πλαίσιο αυτής της ε, προτάσεως. Έχετε από την ανακοίνωση ήδη ενημερωθεί ότι θα υπάρχει δυνατότητα να συζητήσουμε και να δούμε το θέμα αυτό και ανεπίσημα ε, με τον κύριο Βίλαντ και σε, ένα σύντομο, μια σύντομη δεξίωση με ένα σάντουιτς ε, στο διάλειμμα. Έχουμε λοιπόν μια έκθεση η οποία αυτή την εβδομάδα αύριο θα κριθεί ως προς τη νομική της βάση, ένα πολύ σημαντικό θέμα, με την ψηφοφορία και στο τέλος της εβδομάδας θα απασχολήσει και το Συμβούλιο. Ήταν δηλαδή πολύ συνειδητή η επιλογή της σημερινής ημέρας για την ε, συνεδρίαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, θεωρώντας ότι θα έχει πολύ μεγάλη πρακτική αλλά και ουσιαστική σημασία εγκαίρως εμείς να έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό και να αναλάβουμε στη συνέχεια έχοντα συλλέξει τις ιδέες σας στην περαιτέρω επεξεργασία του επιλέξαμε τη συγκεκριμένη ημέρα. Και τώρα θα παρακαλώ την κυρία Ρόδη Κράτσα να αναλάβει εκ μέρους της Επιτροπής των Γυναικών να μας κάνει την παρουσίαση του εγγράφου εργασίας, το οποίο αποτελεί τη βάση για τη σύνταξη της εκθέσεως. Πρόκειται και ένα έγγραφο εργασία το οποίο έχετε ασφαλώς λάβει και εκθέτει τα διάφορα στήματα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ εκ μέρους της Επιτροπής Γυναικών και ως ε, συνεισηγήτρια του θέματος να χαιρετήσω αυτή την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να ε, εκθέσουμε τις απόψεις μας και να ανταλλάξουμε και απόψεις μαζί με συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι αρχή μας σταθερή ότι η δημοκρατία η ευρωπαϊκή και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας υπηρετείται στα δύο επίπεδα, το ευρωπαϊκό και το εθνικό. Ένα τέτοιο θέμα λοιπόν όπως αυτό που μας απασχολεί σήμερα, το οποίο άπτεται πολλών πτυχών της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη, για τη δικαιοσύνη, για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, για την ισότητα, είναι πολύ σημαντικό να το συζητούμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση αυτή δεν ήλθε ξαφνικά στο πλαίσιο της ατζέντα μας της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η, συμμετοχή των, η ισόρροπη συμμετοχή των δύο φίλων στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων έχει ε, να κάνει με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την ισότητα. Παντού αναφέρεται ότι η ισότητα στην οικονομική ζωή, στην πρόσβαση στην οικονομική διαδικασία και στις αποφάσεις τις οικονομικές είναι απαραίτητη, απαραίτητος πυλώνας της πολιτικής για την ισότητα των φύλων. Επίσης αναφέρεται παντού ότι η ισότητα αυτής της οικονομικές αποφάσεις έχει αποτελέσματα και στην αποτελεσματικότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων ως σύνολο της οικονομίας αλλά και ως ε, ικανότητα, αποτελεσματικότητα και επίδοση των ίδιων των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό το Συμβούλιο ήδη από τη δεκαετία του 90 έχει κάνει συστάσεις προς τα κράτη-μέλη για την ισόρροπη αυτή συμμετοχή. Το λέω, αυτό το επισημαίνω, διότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι η σημερινή πρωτοβουλία της οδηγίας έρχεται από μια διαδικασία που ήδη έχει ξεκινήσει και δεν έχει αποδώσει καρπούς. Το Συμβούλιο κάνει συστάσεις από τη δεκαετία του 90 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ισότητα είναι μέσα το θέμα αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2011 ψήφισε μια έκθεση της οποίας είχα την τιμή να μισηγήτρια ακριβώς ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην καθυστερήσει πια και να φέρει μια νομοθετική πρόταση. Διότι παρατηρήσαμε αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι ότι παρόλες τις πρωτοβουλίες που έχουν παθεί σε κάποια κράτη-μέλη παρόλες τις πρωτοβουλίες που επιχειρήσεις μεγάλες ή μικρές παίρνουν ήδη από μόνες τους για να προωθήσουν το θέμα αυτό της ισόρροπης συμμετοχής, η βελτίωση είναι αφενός πολύ πολύ αργή, αφετέρου ανομοιόμορφη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον κατακαιρματισμό της ενιαίας αγοράς, δεν λειτουργεί παντού ομοιόμορφα η ενιαία αγορά, ούτε ως προς τις ε, ε, πρόσβαση που έχουν ε, τις σχέσεις των επιχειρήσεων με τα νομικά καθεστώτα, ούτε προς την κινητικότητα των στελεχών και τις ευκαιρίες που έχουν τα στελέχη, άνδρες και γυναίκες, να παίξουν ένα ρόλο στην διοίκηση των επιχειρήσεων. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα που είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο ανάπτυξης, λειτουργίας της ενιαίας αγοράς που είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματά της, αξιοποίησης του ταλαντούχου προσωπικού της, που είναι επίσης ένα από τα μεγάλα της πλονεκτήματα στον αγώνα για την ανταγωνιστικότητα, είμαστε σύμφωνοι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να έχει μια νομοθεσία η οποία δίνει ένα κοινό πλαίσιο δράσης για όλα τα κράτη-μέλη. Ε, αισθάνομαι ότι δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, αλλά θα πω δύο-τρία σημεία που είναι πιστεύω πολύ σημαντικά ως χαρακτηριστικά της οδηγίας και τα οποία θα μας βοηθήσουν στη συνέχεια για τη συζήτησή μας. Η οδηγία σέβεται την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε σήμερα που έχουμε εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων με έννοια για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους που έχουν στην νομοθετική διαδικασία. Διότι η, η, η οδηγία δίνει ένα κοινό στόχο για τα κράτη-μέλη να πετύχουν στις επιχειρήσεις τους, τις εισηγμένες, 40% συμμετοχής των γυναικών έως το 2020 και μέχρι το 2018 για τις επιχειρήσεις όπου το κράτος είναι, έχει την πλειοψηφία. Δίνει στα κράτη-μέλη το δικαίωμα να εφαρμόσουν μια το δικό τους τρόπο και στις επιχειρήσεις επίσης για να πετύχουν αυτό το στόχο. Ε, δίνει μεγάλη έμφαση σε μια νέα διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει η οποία έχει σχέση με την καλή διακυβέρνηση των επιχειρήσεων που εξασφαλίζει κοινά κριτήρια στην επιλογή και στην εκλογή των υποψηφίων, ε, διαφάνεια στους τρόπους που επιλέγονται οι υποψήφοι, διότι έχουμε διαπιστώσει ότι η έλλειψη κοινών κριτηρίων και διαφάνειας θίγει ιδιαίτερα τις γυναίκες υποψήφιες. Αυτό το πλαίσιο των αρχών και των αξιών της νέας διακυβέρνησης των επιχειρήσεων είναι κοινά μέσω της οδηγίας σε όλα τα κράτη-μέλη, εναπόκειται όμως στις επιχειρήσεις και στα κράτη-μέλη πώς θα εξασφαλίσουν την προάσπιση και την εφαρμογή αυτών των αρχών και των κριτηρίων. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίζουμε αυτό, διότι λαμβάνουμε υπόψη ότι στις διάφορες χώρες μέλη υπάρχουν και διαφορετικά νομικά καθεστώτα ως προς τις επιχειρήσεις και την ε, διοίκησή τους. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Εν ώρα κρίσης δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε με διοικητικές υποχρεώσεις που θα είχαν κόστος στις επιχειρήσεις. Γι' αυτό η οδηγία αναφέρεται στις μη εκτελεστικές θέσεις και δεν υποχρεώνει τη δημιουργία κάποιων ιδιαίτερων δομών μέσα στην επιχείρηση για να υπηρετήσουν αυτό το στόχο. Ε, ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το επισημάνουμε και ε, πιστεύουμε ότι η εφαρμογή αυτή της οδηγίας δεν επηρεάζει τα κράτη-μέλη που έχουν ήδη μια νομοθεσία και έρχεται απλά ως χορηγός στα κράτη και στις επιχειρήσεις που ήδη έχουν επιλέξει να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένο στόχο προώθησης της ισότητας στις, ε, στα κέντρα που λαμβάνονται οικονομικές αποφάσεις. Αυτά τα κράτη-μέλη και αυτές οι επιχειρήσεις ε, ε, δεν έχουν κάτι που είναι αντίθετο προς την οδηγία, απλά η οδηγία δίνει ένα συμπληρωματικό πλαίσιο. Είναι δηλαδή η οδηγία ένα, μια υποχρεωτική ε, ε, υποχρεωτικός στόχος, μια υποχρεωτική διαδικασία για την προώθηση της ε, ισότητας στα κέντρα που λαμβάνονται αποφάσεις. Για τις επιχειρήσεις και για τα κράτη-μέλη που υποστηρίζουν αυτό το στόχο ειλικρινά και θέλουν να έχουν ένα αποτέλεσμα, η οδηγία γίνεται ένα εργαλείο προς την προώθηση αυτού του στόχου. Ε, από την έρευνα που έχω κάνει για την παρούσα οδηγία, για την έκθεση που έχει ήδη ε, ε, ψηφιστεί εδώ και δύο χρόνια, είμαι πεπισμένη ότι μόνο τα κράτη-μέλη τα οποία δεν δίνουν σημασία στην αρχή και στην αξία της ισότητας στα κέντρα που λαμβάνονται οικονομικές αποφάσεις μπορεί να έχουν αντίθεση με την οδηγία. γιατί η οδηγία τους δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσουν και το χρονοδιάγραμμά τους μέχρι το 2020 και τα μέτρα τα οποία αυτά νομίζουν ότι πρέπει να πάρουν για να πετύχουν το στόχο. Είναι δηλαδή ένα θέμα αξιολόγησης της σημασίας της ισότητας, της δικαιοσύνης και της διαφάνειας και δέσμευσης να υπηρετήσουμε το στόχο ε, αυτές τις αρχές θέλουμε να υποστηρίξουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλουμε η αξιοκρατία να επικρατήσει, η διαφάνεια και τα κριτήρια υπηρετούν την αξιοκρατία για άντρες και γυναίκες και να δώσουμε μια όθηση στις γυναικείες υποψηφιότητες ε, που μέχρι σήμερα οι συνθήκες δεν τους το έχουν ε, δεν, τους το έχουν προσφέρει. Στόχος μας δεν είναι οι γυναίκες που δεν θέλουν ή που δεν είναι ικανές να βρεθούν στα κέντρα ε, των να βρεθούν στα διοικητικά συμβούλια. Στόχος μας είναι οι άξιες γυναίκες που, έχουν, ε, πληρούν τα κριτήρια, που έχουν τη φιλοδοξία και το στόχο να βρεθούν στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων να μην συναντήσουν τα εμπόδια που συναντούν σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και για την, ε, Παρουσίασα σήμερα εδώ και είμαι σίγουρη ότι στη συζήτηση θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε ε, θέματα που άπτονται ιδιαίτερων ε, πτυχών της οδηγίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κρέτσα. Θα δώσω τώρα το λόγο σε άλλη συνεισηγήτρια, στην ε, κυρία Ρέγνερ από την πλευρά της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Παρακαλώ αυτή το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πριν να ε, αναλάβω τον ρόλο μου ως συνεισηγήτριας, θα ήθελα πολύ σύντομα, μια και ξεκινήσαμε τόσο, μπήκαμε τόσο άμεσα στο θέμα, θα ήθελα να πω πιο πρακτικά ζητήματα, ότι βλέπετε από το πρόγραμμα είναι εξή εξέλιξη της συζητήσεω. Η κυρία Κράτσα θα παρουσιάζει το ένα κομμάτι του εγγράφου εργασία, το οποίο στη συνέχεια εκβάλλει σε μια έκθεση, το οποίο και, εγώ από πλευράς μου συμπληρώνω. Μετά οι συντάκτριες γνωμοδοτήσεων από άλλες επιτροπές, οι οποίες επίσης θα μιλήσουν, γιατί έχουν τις γνωμοδοτήσεις τους, θα ε, λάβουν το λόγο και στη συνέχεια και εσείς αγαπητοί, αγαπητές βουλευτές από 10 κράτη-μέλη μπορείτε να μας κάνετε τις παρουσιάσεις σας για την κατάσταση σε εθνικό επίπεδο και έτσι θα ολοκληρωθεί η συζήτηση. Πάνω απ' όλα λοιπόν θέλουμε χάρη στη συνεδρίαση αυτή να συλλέξουμε αυτές τις θέσεις για να έχουμε μια πλήρη επισκόπηση της δουλειάς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο βέβαια που θα παρουσιάσουμε εμείς αλλά και των εθνικών θέσεων που θα παρουσιαστούν από πλευρά σα για να μπορέσουμε να τις συζητήσουμε μετά από κοινού. Για το δικό μου λοιπόν τμήμα, για να συμπληρώσω εγώ το δικό μου κομμάτι. Καταρχάς, ε, στη νομική βάση, όπως είπα και στην αρχή, αύριο γίνεται η ψηφοφορία για τη νομική βάση στην Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων, η σχετική με τη νομική βάση. Αρμόδια για τι νομικέ βάσει όπω είναι αρρωστολογικό, είναι η Νομική Επιτροπή και την ψηφίζει ε, υπάρχει μία πρόταση για το άρθρο 157.3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την πρόταση αυτή εγώ θεωρώ ότι είναι ε, κατάλληλη η νομική βάση γιατί έχουμε να κάνουμε την πρόσβαση και όχι με την πραγματική συμμετοχή. Η πρόσβαση λοιπόν για μένα είναι ε, ευφυής, είναι καλά ισορροπημένη και μπορεί να βοηθήσει την πρόοδο της διαδικασία αυτής. Άρα είμαι σύμφωνη με την νομική βάση, αύριο γίνεται η ψηφοφορία. Ως προς την ουσία τώρα και το περιεχόμενο. Ε, σημείο φετηρία είναι, όπως είπε η κυρία Κράτσα, ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου το ποσοστό της, του λιγότερου εκπροσωπουμένου φύλου, για να το πω ξεκάθαρα, των γυναικών, έχει πολύ, ε, πολύ περιορισμένη παρουσία, ενώ ήδη από τις αρχές της σύσταση Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση από τις πρώτες συνθήκες είναι ξεκάθαρα προσδιορισμένος ο στόχος στις συνθήκες της ίσης ε, μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Από τις απαρχές λοιπόν της Ευρωπαϊκής ε, Κοινότητας και Ένωσης υπάρχει δεδηλωμένος αυτός ο στόχος. Αν κοιτάξουμε την κατάσταση στα κράτη-μέλη πάντως, φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει προβλέψει μια σειρά κανόνων comply, explain, ε, με θελοντική δέσμευση, ένα είδος καρότου θα λέγαμε, το οποίο ε, τίνει ενώπιον της μύτης των κρατών μελών να τα πείσει, να προχωρήσουν προς την κατάσταση, προς την τάση αυτή, προς το στόχο αυτό, αλλά δεν τα έχει ακόμη καταφέρει. Και έτσι Κοιτάμε καταρχάς τα κράτη εκείνα στα οποία ε, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, παλιά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι και συνδυάζονται αυτοί οι στόχοι με κυρώσεις, την κατάσταση ώστε να καταγράψουμε καταρχάς και όντως διαπιστώνεται μία πρόοδος. Υπάρχουν και άλλα κράτη τα οποία έχουν εισαγάγει βέβαια κάποια μέτρα με λιγότερο ή περισσότερο δεσμευτικό χαρακτήρα. Στο έγγραφο εργασίας τώρα, συνεχίζω, προτείνουμε να εξεταστεί πιο προσεκτικά το πεδίο εφαρμογής, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περιορίσει το πεδίο εφαρμογής στις εισηγμένες ε, εταιρείε. Ουσιαστικά πρόκειται για τις μεγάλες δηλαδή επιχειρήσεις. Και τίφτε το ζήτημα μήπως θα ήταν ευφιέστερο να στραφούμε και προς μικρότερες επιχειρήσεις εισηγμένες ε, στο χρηματιστήριο, ώστε να τις περιλάβουμε και αυτές. Έστω και αν δεν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εγώ ως Αυστριακή μπορώ να σας πω ότι όταν μιλώ για επιχειρήσεις ε, τέτοιες, μιλώ για 10-20 ε, εργαζομένους. Έστω και αν υπάρχουν μέχρι 250 εργαζόμενοι στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και ως εκ τούτου μπορεί να, προβλέπετε, να αντιστοιχεί αυτό σε μεγάλο κύκλο εργασιών σχετικά. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε και αυτές να τις λάβουμε υπόψη. Και νομίζω ότι μπορούμε να τις, να τις περιλάβουμε. Ένα άλλο σημείο, πόσο δεσμευτικά θα είναι τα μέτρα, ο βαθμός του, της υποχρέωσης που θα προκύπτει. Βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη για βελτίωση της κατάστασης εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διερωτώμεθα αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα διαφανές, καλό, ισορροπημένο σύστημα για την επιλογή των μελών αυτών να επιτύχει το στόχο ή αν τυχόν θα πρέπει και να οριστεί συγκεκριμένη ποσόστηση. Ένα 40% της στόχος φιλόδοξος, ο οποίος θα μπορούσε και αυτός να συμπεριληφθεί στο διατακτικό Και ένα τρίτο μεγάλο πλέγμα, ε, προβληματισμών που θα πρέπει να συζητήσουμε είναι οι κυρώσεις. Μόλις το ανέφερα ότι τα κράτη που έχουν εισαγάγει σύστημα δεσμευτικό με ε, αποτελεσματικές κυρώσεις ε, όπως επί παραδείγματι πολύ υψηλέ χρηματικέ ε, ε, χρηματικές στην Ιταλία σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι σχετικές ε, διατάξεις ή αποκλεισμό από την αποζημίωση για συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια προβλέπεται στη Γαλλία. θα προτείναμε λοιπόν να εξεταστεί αυτό και να κοιτάξουμε την δυνατότητα να στοχεύσουμε το, στο αποτέλεσμα αυτό με μια δημόσια προκήρυξη, γιατί αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για υλοποίηση του στόχου της συμπλήρωσης και με γυναίκες ε, του αριθμού των μη εκτελεστικών μελών στα διοικητικά συμβούλια. Αυτές είναι κάποιες σκέψεις. Θα πρέπει να δούμε βεβαίως ποιο βαθμό θέλουμε να πιέσουμε, μέχρι πού μπορούμε να πιέσουμε και βέβαια για το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να συζητήσουμε γιατί συζητούμε και προγραμματίζουμε τώρα ενώ πρόκειται η ψηφοφορία να γίνει το φθινόμπορο πρώτα στις Επιτροπές μετά στην Ολομέλεια και καθώς πρόκειται για έναν πολύ ευρύ στόχο θέλουμε ασφαλώς ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε αυτή την περίοδο την νομοθετική, σε αυτή τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και ε, θα σας επισημάνω ότι έχουμε πέραν των πολιτικών φραγμών, των φραγμών των πολιτικών ομάδων, συμφωνία, συνένεση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, υψηλές φιλοδοξίες για ένα καλό αποτέλεσμα. Η συζήτηση λοιπόν και με εσά, βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων, πιστεύουμε ότι είναι πολύ κρίσιμη και γι' αυτό σας καλούμε και εσείς να τοποθετηθείτε. Σας ευχαριστώ κύριε Ρέγκνερ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να τοποθετηθεί σχετικά με το ζήτημα αυτό. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ. Καταρχήν, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γυναικών και την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για την οργάνωση αυτού του διαλόγου μεταξύ των νομοθετών και με τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και ευχαριστώ και τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια που δέχτηκαν να παρευρεθούν εδώ σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια άμεση γραμμή επικοινωνίας ε, με τα Εθνικά Κοινοβούλια και για το ζήτημα αυτό. Δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω τις δύο συγγήτριες, ε, την κυρία Κράτσα και την κυρία Ρέγνερ, για την ε, ρεαλιστική προσέγγιση που ακολούθησαν κατά την ε, κατάρτιση των ε, γράφων. Για αυτή την νομοθετική πρόταση που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του περασμένου έτους. Δεδομένου του ότι η πρόταση αυτή ήδη έχει κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και πάνω από 6 μήνες. Δεν ε, χρειάζεται λεπτομέρης ε, παρουσίαση του περιεχομένου της πρότασης αυτής από την πλευρά της Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά θέλω να τονίσω και ακριβώς επειδή συζητούμε εδώ σήμερα με αξιότιμους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων, θέλω να τονίσω ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της πρότασης οδηγίας. Συγκεκριμένα την έμφαση που δώσαμε στο θέμα της διαφάνειας των κριτηρίων που θα προσδιοριστούν από τους εργοδότες όταν ε, θα επιλέξουν να προσλάβουν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και επίσης ε, για τα διαφανή κριτήρια που ακολουθούνται κατά την επιλογή των μελών των εποπτικών συμβουλίων. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπρος και ένα μεγάλο εμπόδιο που υπήρχε μέχρι τώρα. Δηλαδή γυναίκες με κατάλληλα προσόντα αντιμετώπιζαν αυτό το εμπόδιο. Και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που θέλω να τονίσω ως σημαντικό για αυτή την νομοθετική πρόταση είναι το εξή ότι το σύστημα που προτείναμε σκοπεύει να βασίζεται τα προσόντα αυτών των γυναικών που θα μπουν στα συμβούλια των εταιριών, δηλαδή να λειτουργεί αξιοκρατικά. Και Επομένως, η προτεραιότητα που θα, γίνεται, που θα δίνεται στις γυναίκες δεν θα βασίζεται στο γεγονός ότι είναι γυναίκες. Μιλάμε εδώ για άτομα που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες για να καλύψουν τις θέσεις αυτές. Και επειδή σήμερα εδώ συζητούμε με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, θα ήθελα να παρουσιάσω ορισμένα στοιχεία τα οποία μας δείχνουν τη συμμόρφωση της νομοθετικής μας πρότασης με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Καταρχήν, να επαναλάβω και μία δήλωση που έχει γίνει ήδη εδώ, με δύο λόγια ότι αυτή η ανησυχία για την ισότητα των φύλων και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων και στα Συμβουλία των Εταιριών δεν είναι μια ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ισότητα των δύο φύλων υπάρχει στις ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, αυτό ήδη δίνει ένα, μια μερική απάντηση σε όσους ανησυχούν ε, για την παραβίαση της αρχής της με μέσα στη δυναμοθετική πρόταση. Να προσθέσω ότι παρά το ότι είναι παλιά αυτή η ανησυχία και είναι και παλιά αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ε, περασμένες δεκαετίες, ε, δεν είδαμε να σημειώνεται ιδιαίτερη πρόοδος. Και θα σας παραπέμψω μόνο στα τελευταία δημόσια νούμερα σήμερα έχουμε 15,8% γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια τον Οκτώβριο του 2012 και υπήρξε μια αύξηση το τελευταίο έτος στις περισσότερες χώρες μέλη με εξαίρεση τρία κράτη-μέλη. Τώρα, αυτό μας δείχνει ότι η κατάσταση είναι σχετικά μετριοπαθής, η πρόοδος είναι αργή στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς αξιολογήσαμε και το γεγονός ότι τα σημεία φετήρια σε κάθε κράτος μέλος μπορεί να διαφέρουν. Και επίσης ότι οι λύσεις που βρέθηκαν από διάφορα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού μπορεί να διαφέρουν. Η πρότασή μας έχει συμπεριλάβει ένα χαρακτηριστικό ευελιξίας που καλύπτεται από το άρθρο 8 και επιτρέπει στα κράτη-μέλη που μπορούν να αποδείξουν ότι οι εθνικές τους λύσεις λειτουργούν καλύτερα ή είναι τόσο αποτελεσματικές όσο οι λύσεις που έχουν κατατεθεί από την Κομισιόν, να μπορούν να επιλέξουν τις δικές τους προσωρινές λύσεις, εθνικές λύσεις και προσωρινά να αναστείλουν τις απαιτήσει διαφάνειας που καθορίζονται από την οδηγία αυτή. Να τονίσω επίσης ότι ήδη ελέγξαμε, έγινε έλεγχος της επικουρικότητας από την Εθνικά Κοινοβούλια όταν κατατέθηκε η πρόταση αυτή και το γενικό αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι θετικό. Δηλαδή, ενώ κάποια εθνικά κοινοβούλια τοποθετήθηκαν αρνητικά για τη συμμόρφωση της πρότασης αυτής με την αρχή της επικουρικότητας και είχαμε γραμματοτήσεις από έξι κρατημέλη. Συνολικά το κατόφλι των 18 ε, ψήφων ε, από τις 54 πόρες από τη συνθήκη δεν ε, το επιτεύχθη. Έτσι λοιπόν αυτό δείχνει ότι τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια υποστήριζαν την πρόταση αυτή και θεωρούσαν ότι συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Και για να κλείσω να πω δύο λόγια για τις ανησυχίες σε σχέση με το σεβασμό της αρχής της, της αναλογικότητας. Εμείς πήραμε σοβαρά αυτό το θέμα και αυξήσαμε την ευελιξία της νομοθετικής μας πρότασης ή πολύ συγκεκριμένα στοχεύσαμε στα κύρια θέματα ανησυχίας. Γι' αυτό ακριβώς η πρόταση στοχεύει να καλύψει τα εποπτικά συμβουλία των χωρών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, των εταιριών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, στα κράτη-μέλη μας και όχι τις ε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί πιστεύουμε ότι μεγαλύτερες εταιρείες έχουν καλύτερους και περισσότερους πόρους και καταλληλότερες δομές και είναι πιο ικανές να διαχειριστούν τη διαδικασία της κατάρτισης διαφανών κριτηρίων για τις προσλήψεις. Έτσι λοιπόν μπορούν να προσλάβουν τις ε, ικανές γυναίκες ε, για τα διοικητικά συμβούλια καλύπτουμε εδώ και τα κλειστικά συμβούλια και τα εποπτικά συμβούλια, αλλά με διαφορετικό τρόπο, με έναν τρόπο να δούμε ποιες είναι, να αναγνωρίσουμε αυτές τις διαφορές. Για τα εποπτικά συμβούλια έχουμε προτείνει ένα στόχο 40% των γυναικών μέχρι τα τέλη της σημερινής δεκαετίας. Ήδη αυτό ορίζεται στην οδηγία και θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό μέσω της ε, νομοθεσίας που θα εφαρμοστεί ε, από τα κράτη-μέλη, ενώ για τα εκτελεστικά συμβούλια το έχουμε αφήσει αυτό το θέμα περισσότερο στα χέρια των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων εταιριών. Και η διγεία αποτελεί μόνο από τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν στι εταιρείε δημοσίως να αναλαμβάνουν στόχους για να βελτιώσουν την εκπροσώπηση των δύο φύλων στα εκτελεστικά του συμβούλια. Να τονίσω επίσης ως ένα άλλο στοιχείο που βεβαιώνει την ανησυχία μας για την αναλογικότητα, το ότι δεν έχουμε καταθέσει προς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση που να στοχεύει να εφαρμοστεί μια νομοθεσία επάπειρων. Υπάρχει μια ρήτρα λήξη της ισχύω ε, μεταξύ των διατάξεων και λέει αυτή ότι όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όταν ε, έχουν υλοποιηθεί οι στόχοι θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση βάσει της υποβολής εκθέσεων, βάσει των εκθέσεων που θα υποβληθούν από τα κρατημέλη θα πρέπει να γίνει με τη αξιολόγηση από την Κομισιόν και η εφαρμογή αυτού του νομοθετήματος θα πρέπει να πάυσει. Να κλείσω την παρέμβασή μου. Εκμεταλλευόμαστε στο γνώση ότι έχουμε εδώ εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων σήμερα για το διάλογο αυτό και να απευθύνω μια έκκληση σε αυτούς και να υποστηρίξουν αυτό το ζήτημα στα αντίστοιχα Εθνικά Κοινοβούλια και να συνεχίσουν να δίνουν έμφαση στην ανάγκη να έχουμε μεγαλύτερη ισότητα των δύο φύλων, όχι μόνο στη δημόσια ζωή, αλλά και στην οικονομική ζωή, στις λήψεις αποφάσεων στον οικονομικό τομέα και στη δίκηση των εταιριών. Και να απευθύνω και μια έκκληση σε αυτούς να υποστηρίξουν αυτή την προσέγγιση και την νομοθετική πρόταση που κατατέθηκε από την Κομισιόν στα τέλη του περασμένου έτους ενώπιον των κυβερνήσεών τους, να ασκήσουν πίεση δηλαδή στις κυβερνήσεις τους, να υπάρξει θετική ψήφο στο Συμβούλιο για αυτή την νομοθετική πρόταση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και να δώσω τώρα το λόγο στην εκπρόσωπο του Συμβουλίου, την κυρία Πολύν Μωρό από την Ιρλανδία, την Ιρλανδική Προεδρία. Thank you very much Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε και για την πρόσκληση να παραβρεθούμε στη συζήτηση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό Συμβούλιο και Κοινοβούλιο συνομοθέτες να συνεργαστούν σε όλη αυτή την νομοθετική διαδικασία και χαίρομαι για τις απόψεις που ακούω σήμερα. Η Ιρλανδική Προεδρία αφιέρωσε τέσσερις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας Κοινωνικών Ζητημάτων στο θέμα αυτό. Είχα την τιμή να προεδρεύσω και μπορώ να σας πω πως η συζήτηση συμπεριέλαβε όλα τα κράτη-μέλη. Η συζήτηση στην ομάδα αποκάλυψε πως υπάρχει ευρεία συνένεση υπέρ του βασικού στόχου της πρότασης, δηλαδή να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων των εταιριών στο υψηλότερο επίπεδο. Όμως, οι απόψει αποκλίνουν ε, όσον αφορά τον καλύτερο τρόπο επίτευξη αυτού του στόχου. Κάποιε αντιπροσωπείε υποστήριξαν την προσέγγιση τη Κομισιόν και από αυτέ ε, πολλέ ήδη έχουν αναλάβει δρα... πρωτοβουλίες θετική δράσης που όπω αναφέρθηκε ήδη έχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Από την αξιολόγηση αντικτύπου που προετοίμασε η Κομισιόν, η ομάδα εργασία επίση σημείωσε την έρευνα η οποία αποδεικνύει πω ε, πιο επιτυχημένε είναι οι εταιρείε οι οποίε έχουν σε εκπροσώπηση των φίλων, αλλα Άλλα κράτη-μέλη είχαν την άποψη πως ε, δεν γίνεται σεβαστή η αρχή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Επίσης αμφισβητήθηκε η νομική βάση από λίγες χώρες. Μια άλλη ομάδα χωρών προετοίμασε μια εθελοντική λύση που θα επέτρεπε στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια για να αποφασίσουν τις πολιτικές τους. Η υπερτινόμενη οδηγία προτείνει πως ε, για να επιτευχθεί μεγαλύτερη εκπροσώπηση του υποεκπροσωπούμενου φύλου θα έπρεπε να τεθεί ένας στόχος είτε 40% είτε 33% και για τα εκτελεστικά και μη μέλη του ΔΟΣΟΥ. Και όπως είπαμε και στις συζητήσεις μας κάποια κράτη-μέλη επεσήμαναν πως ξεκινούσαν από μια πάρα πολύ χαμηλή αφετηρία όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στις εταιρείε και σημείωσαν πως η πρόταση της ε, Κομισιόν ε, ήταν μια πραγματική πρόκληση όσον αφορά την επίταξη του 40% μέχρι το 2018, ειδικά μέχρι το 2020 και για το 2018 για τις εισηγμένες. Η ετήσια έκθεση της Κομισιόν δείχνει πως αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 16% και 16 κράτα-μέλη είναι κάτω από αυτό το μέσο όρο. Βεβαίω είναι τεχνικό το θέμα και εδώ πέρα βεβαίω πρέπει να λάβουμε υπόψη διαφορετικές πρακτικές και διαφορετικό εταιρικό δίκαιο. Θα απαιτηθεί λοιπόν περαιτέρω έντονη εξέταση στο επίπεδο ομάδα εργασίας και κρατών μελών. Η μελλοντική εργασία μας λοιπόν επί του θέματος σημαίνει πως ε, συνεργαζόμαστε και με τους Λιθουανούς συναδέλφους και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε ένα κείμενο με τις προτάσεις μας. Αν μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να ευχηθώ στους Λιθουανούς συναδέλφους καλή επιτυχία στη συνέχεια του φακέλου αυτού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Έχουμε και εκπρόσωπο από την επόμενη Λιθουανική Προεδρία του Συμβουλίου. Παρακαλώ, κύριε Κόβα, και έχετε το λόγο. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές ε, του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετάσχω σε αυτή την ενδιαφέρουσα και ζωντανή συζήτηση. Το Συμβούλιο είναι στις πρώτες φάσεις ε, της εξέτασης ε, του φακέλου αυτού και οι προτάσεις διαφέρουν όμως είναι ήδη προφανές πως υπάρχει ευρεία συνένεση μεταξύ των κρατών μελών για την ανάγκη να γίνουν περισσότερα για να αυξηθεί ο αριθμός γυναικών στη λήψη αποφάσεων ειδικά σε επιχειρήσεις. Η Λιθουανία ως μελλοντική προεδρία θα συνεχίσει βεβαίως ε, τις συζητήσεις με τους συνεργάτες μας στην ε, τριπλή προεδρία οι συζητήσεις δεν θα είναι εύκολες, βλέπουμε όμως κάποιες δυνατότητες να υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση σε κάποια εκκρεμή ζητήματα που ανέφεραν οι συνάδελφοι από την Κομισιόν και την Τρέχουσα Προεδρία που πρέπει βεβαίως ακόμα να λυθούν για να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια στις προτάσεις. Ειδικά το πεδίο εφαρμογής, η διάκριση μεταξύ διαδικασιών επιλογής και προεπιλογής, ε, δημοσιοποίηση πληροφοριών και κυρώσεις. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε πως το σχέδιο οδηγίας ε, εμπεριέχει αρκετή ευελιξία και επιτρέπει στα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες όταν θα εφαρμόσουν την οδηγία. Σέβεται την ποικιλομορφία που υπάρχει ε, όσον αφορά το εταιρικό δίκαιο και τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί για να βελτιώσουν τη θέση των γυναικών. Η πτυχή αυτή πρέπει να συζητηθεί επίσης και να ξεκαθαρίσει. Τέλος, η Λιθανική Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να προχωρήσει το θέμα αυτό στο επίπεδο του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Νόβακ. Και τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων και φυσικά και τους ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του Συμβουλίου που δεν μακρηγόρησαν για να μπορέσουν να επιτρέψουν σε όλους ε, να πάρουν το λόγο, σε όλους όσους το επιθυμούν δηλαδή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, γιατί και οι συγγήτριες θέλουν να ακούσουν τις δικές σας ιδέες και προτάσεις που ενδεχομένως θα συμπεριλάβουν στην εκθεσή τους. Μια πρώτη ομιλήτρια έχουμε από το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας. Έχετε το λόγο, όμως θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σεβαστείτε τα τρία λεπτά της παρέμβασής σας. you so much. Good morning. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την ε, ευκαιρία να παρευρεθώ εδώ σήμερα το πρωί και να υποστηρίξω την ιδέα της εκπροσώπησης, ε, της ισορροπημένης εκπροσώπησης των δύο στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών ε, και να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας για το θέμα τη ισότητα των δύο φύλων στη Λιθουανία. Η ισότητα των δύο φύλων και εσείς ευκαιρίε είναι θεμελιώδη στο όχι που προσπαθεί να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως ε, συνεχίζει να υπάρχει διερημένη υποστήριξη στα κράτη-μέλη, καθώ οι πολιτικοί στις ε, εθνικέ κυβερνήσει και κοινοβουλία έχουν αποκλίνουσες ε, πολιτικές απόψεις και εκπαιδευτικό background. Η κατάσταση στη Λιθουανία είναι παράδοξη, καθώ η ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών χαρακτηρίζονται περισσότερο από προοδευτικό σκεπτικό στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων, από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μία δημοσκόπηση που έγινε το 2011 μας δείχνει ότι το 89% των Λιθουανών πολιτών συμφωνούν να υπάρχει ίση εκπροσώπηση ενδρών και γυναικών στις διοικητικές θέσεις της επιχειρήσης οι απαντήσεις ήταν ε, ε, διαφορετικές σε σχέση με το πώς θα το πετύχουμε αυτό. 27% υποστήριζαν την νομοθεσία, ενώ 27% τη ρύθμιση της επιχειρήσης, 27% υποστήριζαν δεσμευτικά νομοθετικά μέτρα και άλλοι υποστήριξαν εκούσιες πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων. Όμως η πλειοψηφία, το 78% θα υποστήριζε νομικά δεσμευτικά μέτρα, δίνοντας προτίμηση στα προσόντα και στις δεξιότητες, ε, παρά ε, στην αυτόματη εφαρμογή της επιλογής βάσει του φύλου. Και ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητούσε την πρόταση για τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις για τις γυναίκες ε, στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών, των συγμένων εταιριών, απουσία συγκεκριμένων ε, προτάσεων, οκτώ κράτη-μέλη και η Λιθουανία προσέβαλαν την, από, την ε, πρόταση και εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην υιοθέτηση οποιονδήποτε δεσμευτικών ευρωπαϊκών διατάξεων για το θέμα των ποσοστών των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Τότε ο Λιθουανός ε, Υπουργός ε, ε, Εργασίας ανήκε στο Συντηρητικό Κόμμα. Όμως αφού η Κομισιόν κατέθεσε την πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της εκπροσώπησης των δύο φύλων μεταξύ των μη ε, εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων ε, στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. Ε, υπήρξε μια τροποποίηση. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αξιολογήθηκε από άτομα ναι, που είχαν αναλάβει τα καθήκοντά τους και επίσης ήθελαν να προωθήσουν την συμμεταχείριση ανδρών και γυναικών, αλλά διερωτήθηκαν αν το επιχείρημα της Κομισιόν σε σχέση με την έλλειψη πρωτοβουλίας ε, από τα κράτη-μέλη αιτιολογούσε την ανάγκη αντίδραση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή αποφάσισε πως η πρόταση ίσως να είναι σε αντίθεση με την αρχή της επικουρικότητας. Σε αυτή την θητεία η Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελείται κυρίως από συντηρητικούς βουλευτές που μερικές φορές χρησιμοποιούν ε, κάποιες τεκαλυμμένες φράσεις για να καλύψουν ε, αυτό το ζήτημα. Επίσης και η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συζήτησε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το αν σέβεται την αρχή της επικουρικότητας. Υπήρξαν πολλές ακροάσεις για την πρόταση αυτή. Εγώ ήμουν ε, ένα από τα μέλη της Επιτροπής, αρμόδια να συντάξω τα συμπεράσματα και έπρεπε να επενθυμίσω στην Επιτροπή ε, το ιστορικό της ανισότητας των δύο φύλων ε, για να τονίσω τη θετική διάκριση ως απαραίτητο μέσο να πετύχουμε την ισότητα των δύο φύλων στην κοινωνία, καθώς και τα θετικά αποτελέσματα και την αποτελεσματική συνεισφορά των γυναικών στην οικονομία. Με μετά από μια έντονη συζήτηση για το θέμα των ποσοστώσεων, οι ψήφοι από τους σοσιαλδημοκράτες καθόρισαν την απόφαση της ε, Επιτροπής ότι σέβεται, δηλαδή την αρχή της επικουρικότητας ε, η οδηγία. Η οι πολίτες ε, τώρα που είναι αντίθετοι θεωρούν ότι οι ποσοστώσεις εξευτελίζουν τις γυναίκες ε, τονίζοντας ε, την νοητική τους κατωτερότητα. Όλες οι εξηγήσει για την απόρριψη των ποσοστώσεων προκύπτουν από την άγνοια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν τους λόγους των διακρίσεων κατά των γυναικών και πολλοί πιστεύουν ότι σε μια χώρα που διαφυλάσσει τις παραδοσιακές οικογενειακές αξίες, οι γυναίκες ε, που επιθυμούν ε, τη βελτίωση της ε, σταδιοδρομία τους ουσιαστικά δεν επιδεικνύει αλληλεγγύη στους άνδρες δεν βλέπουμε ενοποιημένες στρατηγικές δράσεις να υπερασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δημιουργούν πολιτικές ισότητες των δύο φύλων σε κυβερνητικό επίπεδο στη Λιθουανία. Η έλλειψη δράση στην πρόθεση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ισότητας των δύο φύλων από την κυβέρνηση τονίστηκε πρόσφατα στην έκθεση του Human Rights Watch που επίσης προειδοποίησε ότι η... στη λιθουανική κοινωνία επιδεινώνεται η κατάσταση σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε κρατικό επίπεδο υπάρξει, υπάρχει έλλειψη υποστήριξη για νέε πτυχέ ισότητα των δύο φύλων. Οι προτάσει από το γραφείο του διαμεσολαβητή για την ισότητα των δύο φύλων δεν λαμβάνονται υπόψη από την κυβέρνηση πολύ λίγα μέλη του Κοινοβουλίου αγωνίζονται για νέες τροπολογίες, για τροποποίηση της νομοθεσίας, για τις ίσες ευκαιρίες. Το πρόγραμμα του Συλλοδημοκρατικού Κόμματος της Λιθουανίας υπογραμμίζει την ισότητα των δύο φύλων και των ίσων ευκαιριών. Είναι το μόνο κόμμα στη Λιθουανία που έχει εισαγάγει ποσοστώσεις για τους υποψηφίους τους εκλογές. αυτή η απόπειρα εισαγωγής ε, ποσοστώσεων για τις γυναίκες απέτυχε το 2003 και το 2011 όταν περίπτω τη δισάιτεν ε, συνέταξε ένα νομοσχέδιο για ίσες ευκαιρίες για τους άνδρες και τις γυναίκες που πρότεινε στις τοπικές αρχές και στις κρατικές αρχές να διασφαλίσουν ότι το 30% ε, των ανώτερων θέσεων στις εταιρείες ε, καλύπτονται από γυναίκες. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία αντιτάχθηκε και στα δύο νομοσχέδια και μάλιστα απέριψε την πρόταση τροποποίησης του νομοσχεδίου. Συνοψίζοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι πάρα πολλά πρέπει να γίνουν στη Λιθουανία για την πολιτική ισότητα των δύο φύλων, αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι τα προοδευτικά μέλη του Κοινοβουλίου υποστηρίζουν ένθερμα την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ισορροπή εκπροσώπηση των φύλων στις εταιρείε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Παύλη και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Βίρο Λάιναν από τη Φινλανδία. Κυρία Λάιναν, πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω την ε, μητρική μου γλώσσα. Κυρία Πρόεδρε, η Φινλανδία τάσεται υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι και ευθυγραμμισμένη με το πρόγραμμα της Φινλανδικής κυβέρνησης, που επιδιώκει την πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και έχουμε μέτρα ήδη στη Φινλανδία από την κυβέρνηση, αλλά και εθελοντικά μέτρα που έχουν εισαγάγει ήδη στις φιλανδικές επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν έχουμε στη θέση μας τα κατάλληλα εργαλεία για να βελτιώσουμε την ισότητα των φύλων. Στη Φινλανδία μέχρι τώρα έχουμε εισαγάγει ποσοστώσεις εδώ και αρκετό καιρό. Χρόνια πριν κάποιες από τις πρώτες ποσοστώσεις και έτσι έχουμε 40% του λιγότερο εκπροσωπημένου φύλου ως υποχρεωτική συμμετοχή, ως ποσόστος δηλαδή. Αλλά δεν έχουμε δει ουσιαστικέ βελτιώσεις. Το 2005 ήμουν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, εγώ προσωπικός, στην ε, ιδιαίτερη πατρίδα μου, ε, στις εταιρείε που υπάγονται στο δημόσιο ή που ανήκουν στο κράτος. Ε, έχουμε αντίστοιχη υποεκπροσώπηση. Και έτσι θα πρέπει να κοιτάξουμε και σε σχέση με αυτές τη δυνατότητα για ε, επίτευξη της ποσότητας του 40%. Έχουμε ένα ποσοστό μόνο 27 εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών διευθυντών ε, γυναίκες και πάλι και στα υπόλοιπα ποσοστά, ε, στις υπόλοιπες αστικές είναι χαμηλότερο από το 40% το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην διοίκηση των επιχειρήσεων. Ε, άρα λοιπόν, ναι, υπάρχει νομοθεσία στη Φιλανδία, επιδιώκουμε την ε, ίση εκπροσώπηση, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο στόχο αυτό ακόμα. Και θέλουμε να επιτύχουμε το 40% για τις εταιρείες της συγκεκριμένες στο χρηματιστήριο, ε, το 2014 είναι για μας ένας, ε, ένα ορόσημο, διότι εάν δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τότε το επιδιωκόμενο ποσοστό θα εισαχθεί νέα νομοθεσία. Έχουμε για τις συγμένες επιχειρήσεις 23% μόνο συμμετοχή των γυναικών. Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις όμως από τις εισηγμένες έχουμε φτάσει μέχρι το 31%. Είναι υψηλότερο το ποσοστό. Στους ε, εσωτερικούς κανονισμούς διαχείρισης των επιχειρήσεων υπάρχει αναφορά στην ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Ε, ήδη λοιπόν υλοποιείται αυτός ο στόχος της εθελοντικής της αυτοδέσμευσης και η Φιλανδία πιστεύω ότι είναι μια χώρα καλή για τις ευκαιρίες, καταρχάς γιατί είναι πολύ ισότιμη και ισόρροπη η εκπαίδευση μεταξύ των δύο φίλων Είναι πάρα πολύ καλές οι συνθήκες μέρημνας για τα παιδιά, γιατί τους προσφέρεται στο σχολείο το δωρεάν γεύμα, γιατί υπάρχει φροντίδα ή φύλαξη για τα παιδιά, γιατί είναι ε, γιατί μοιράζονται τα άνδρες και γυναίκες τα βάρη της φροντίδας των παιδιών και Όπως είπαμε, εάν δεν βελτιωθεί η κατάσταση ως προς τις ε, εισηγμένες επιχειρήσεις, θα χρειαστεί να εισαχθεί νέα νομοθεσία, αλλά προτιμούμε περισσότερο να δίνουμε κίνητρα παρά κυρώσεις. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Βερόνια Κάθλιν από το Βουλή των Λόρδων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση και μπορούμε να ανταλλάξουμε πληροφορίες ε, και για το τι γίνεται στις χώρες μας, αλλά και να ακούσουμε τα διάφορα επιχειρήματα. Εγώ είμαι πρόεδρος ε, της Επιτροπής ε, της Βουλής των Λόρδων με αρμοδιότητα για την εσωτερική αγορά, υποδομές ε, και απασχόληση και σήμερα θα μιλήσω από σκοπιά της απασχόλησης, αν και βεβαίως έχει τεράστια σημασία η ισότητα των φύλων και για την εσωτερική αγορά. Πέρυσι τον Νοέμβριο η Επιτροπή μας δημοσίευσε μία έκθεση που λεγόταν Women on Board, τρεις μέρες δηλαδή πριν βγάλει την ε, οδηγία η Κομισιόν και ήταν αποτέλεσμα έρευνα στο ζήτημα της ε, ισορροπίας των δύο φύλων στα διοικητικά συμβούλια υπάρχουν στο site μας αυτά. Και μας προξένησε, μας προξένησε έκπληξη ο ε, χαμηλός αριθμός γυναικών στα διοικητικά συμβούλια στην Βρετανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει σημειωθεί πρόοδος. Και εγώ είχα εμπειρία από διοικητικά συμβούλια. Ήμουν σε διοικητικά συμβούλια 6 εταιριών του δίκτυ των Financial Times, των 100 μεγαλύτερων εταιριών, όχι ταυτόχρονα, σε 6 εταιρείε. Και τότε οι γυναίκε ήταν 0,4% ήταν προετών. Αλλά βεβαίω έχει σημειωθεί πρόοδο. Παρ' όλα αυτά, αν δούμε τα γεγονότα, παραδείγματος χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο οι γυναίκε είναι 45% των εργαζομένων, 60% των αποφύτων πανεπιστημίου και δεν είναι δυνατόν να είναι μόνο 17% των ε, μελών ε, των 100 μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών. Αν και σήμερα συνειδητοποιώ πως είμαστε τουλάχιστον στις τρει καλύτερε χώρε. Είμαστε πάνω από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Κράμφιλντ επιβεβαιώνει πω. Υπάρχουν πολλές γυναίκες με τις ικανότητες για αυτές τις θέσεις και ανέφερε 2.500 γυναίκες που θεωρούνται έτοιμες για δοσού. Παράλληλα, οι ε, ευρωπαϊκές ε, σχολές διοίκησης επιχειρήσεων ε, έχουν καταρτήσει καταλόγους με χιλιάδες γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό καθιστά σαφές πως τα ωφέλη για τις επιχειρήσεις και τις γυναίκες θα είναι μεγάλα. Οπότε συμφωνούμε απολύτως με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο είναι δύσκολο είναι ε, άμεση σύνδεση με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Αλλά το ερευνούμε και αν μπορέσουμε να το αποδείξουμε νομίζω πως θα, θα είναι ένα καταιγιστικό επιχείρημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως δραστηριοποιείται στο ζήτημα της σότα σε όλα τα επίπεδα και στα διοικητικά συμβούλια και αυτό το έχει πει και η Επίτροπος Ρέντινγκ. Εμείς προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ένα ηγετικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας και στην έκθεσή μας λέμε πώς θα πρέπει η Κομισιόν να δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και να αξιολογήσει το πόσο καλά αντιμετωπίζουν το ζήτημα τα κράτη-μέλη. Και ενώ υπάρχει σαφής ρόλος για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό, ανησυχούμε για τις ποσοστώσεις ως μέσο. Θεωρούμε πως ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ποσοστώσεις μόνο όταν δεν επιδεικνύουν διάθεση αλλαγή ή κάτι το οποίο δεν ισχύει. Και την Δευτέρα μάλιστα, σε μια ερέτηση στη Βουλή των Λόρδων, ε, κατονομάστηκε μια εταιρεία από τις 100 μεγαλύτερες ε, στο χρηματιστήριο του Λονδίνου γιατί δεν είχε γυναίκες ε, στο δουσού και φαντάζομαι ότι τις επόμενες μήνες θα αλλάξει στάση. Οπότε αυτό το οποίο κοιτάμε είναι κάτι το πιο βιώσιμο από τις ποσοστώσεις. Δηλαδή καλό είναι για τα στατιστικά στοιχεία αλλά δεν αντιμετωπίζονται οι αιτίε της ανισότητας των φύλων. Δηλαδή το ότι δεν πηγαίνουν γυναίκες στις ανώτερες θέσεις της διοίκησης. Και επιπλέον βλέπουμε πως και αρκετές γυναίκες δεν το θέλουν καθώς ε, κινδυνεύει να υπάρξει η αντίληψη πως οι γυναίκες δεν βρίσκονται στα δοσούμε βάση την αξία τους. Ανησυχούμε για το ότι δεν γίνεται σεβαστή επίσης η αρχή της επικουρικότητας που αναφέρεται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, δηλαδή ότι και τα πράγματα πρέπει να γίνονται στο εθνικό επίπεδο, εκτός εάν μπορούν να γίνουν καλύτερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ πέρα δεν λαμβάνεται υπόψη το γενικότερο πλαίσιο, ο ρυθμός της αλλαγής, ακόμα και η ονοματολογία. Εμείς δεν έχουμε εποπτικά συμβούλια, οπότε υπάρχει ένα ζήτημα. Εδώ πέρα υπάρχουν και πολιτισμικές θα διαφορές. Δεν ε, έχουμε πιστεί επίσης για την αναγκαιότητα του 40% αντί για το 30% που λέγαμε παραδοσιακά. Το σκεπτικό εδώ πέρα είναι πως ε, το 40% θα διασφαλίσει μια κρίσιμη μάζα. Εδώ πέρα δεν λαμβάνεται υπόψη ε, δεν λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές δομές στο κάθε κράτος μέλος και ιδιαίτερες απαιτήσει ε, του κάθε δουσου, εάν είναι τεχνική η φύση της εταιρείας κτλ. Επίσης ε, υπάρχει ένας σαφής ρόλος για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει την ισότητα των ε, δύο με άλλα μέση. Ένας, ε, ένα τέτοιο μέσο είναι οι βέλτιστες πρακτικές. Κατά τη διάρκεια της ερευνάς μας είδαμε πως πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, είχαν ενσωματώσει τέτοιες απαιτήσει στους κώδικες εταιρικής διαίκησης και αυτό ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα συμπεριλαμβάνεται και μια διακήρυξη της πολιτικής των δουσού όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί εδώ πέρα να εκδώσει μια μη δεσμευτική σύσταση που θα προτείνει βεβαίως κάποια στιβαρή ε, δράση αλλά και θα έχει τη δυνατότητα να κινητοποιηθεί σύμφωνα με τις συνθήκες όταν τα κράτη-μέλη δεν ε, αναλαμβάνουν δράση. Τέλος, όσον αφορά το μέλλον, προσωπικά πιστεύω πως θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη να κοιτάξουν πέρα από τα νούμερα των γυναικών και να επισημάνουν νεαρές φιλόδοξες γυναίκες και να ανοίξουν το δρόμο τους για τις ηγετικέ θέσεις και νομίζω πως αυτό θα είναι υποφελές για όλους και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Βαρόνη. Θα δώσω τώρα το λόγο στο πρώτο ευρωβουλευτή που έχει δει το λόγο, υπενθυμίζοντας για μια ακόμη φορά πως πρέπει να σεβαστείτε το χρόνο ομιλίας. Μόνο τρία λεπτά σας παρακαλώ. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουν όλοι όσοι το επιθυμούν να πάρουν το λόγο. Η κυρία Κορνέλισεν είναι αρμόδια για την γνωμοδότηση ε, της Επιτροπής Απασχόλησης για αυτό το ζήτημα και επομένως ε, θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Κορνέλισεν και φυσικά είναι και μέλος ε, της Επιτροπής Γυναικών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους εκπροσώπους ε, των Εθνικών που βρίσκονται εδώ για να συζητήσουν αυτό το θέμα μαζί μας. Ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε από κοινού για να καταλήξουμε σε μια καλή οδηγία που να μπορεί να είναι αποδεκτή σε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη-μέλη ή τουλάχιστον όσο χρειάζεται για να περάσει από το Συμβούλιο. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμη κάποιος φόβος ε, γύρω από αυτήν την οδηγία και εγώ δεν το θεωρώ απαραίτητο. Ίσως ε, θα ήταν καλό να το έχουμε κατά νου. Εδώ μιλάμε μόνο για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες και για τις μη εκτελεστικές εταιρείες διοικητικές θέσεις και αυτό σημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής δεν είναι και τόσο ευρύ. Εγώ προσωπικά ίσως θα προτιμούσα διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, ε, αλλά θα ε, προτιμούσα μια πιο στενή οδηγία, δηλαδή καλύτερα να έχουμε μια πιο στενή οδηγία που θα εφαρμοστεί παρά μια ευρύτερη που δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Αυτό σημαίνει, παραδείγματο χάρη, από στοιχεία που έχουμε στη Λουβικία, έχουμε μόνο ε, έχουμε συμμόρφωση, μιλάμε για 28 γυναίκες μόνο που πρέπει να διοριστούν ακόμη. Τώρα, εμείς στην Επιτροπή Επασχόλησης τι προσπαθήσαμε να κάνουμε στην γνωμοδότησή μας, να πλουστεύσουμε την οδηγία έτσι όπως προτείνεται από την Κομισιόν, έτσι ώστε να λέει ότι πρέπει ή να συμμορφωθεί σε να εξηγήσει και αν όχι θα επιβληθούν κυρώσει. Επίση, ε, ενδυναμώσαμε τη δυνατότητα των κρατών μελών να ζητήσουν αναστολή αν ήδη έχουν πολιτικές σε εθνικό επίπεδο, ακόμη και αν είναι εκούσιο χαρακτήρα οι πολιτικές αυτές, τα κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα. Στη Βρετανία θα μπορούσατε να ζητήσετε εσείς αυτή την αναστολή, το ίδιο ισχύει και για τη Φιλανδία τότε το 2017 θα γίνει μια αξιολόγηση και αν έχει σημειωθεί η απαιτούμενη πρόοδος, θα επεκταθεί και η αναστολή. Για τις εταιρείε που συμμορφούνται ή που σημειώνουν την κατάλληλη πρόοδο, θα έχουν πολύ ελαφρές υποχρεώσεις, σύμφωνα με αυτά που προτείναμε εμείς, υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Επομένως, ε, όταν ε, λειτουργούν τα πράγματα, ούτε καν θα προσέξουν ότι υπάρχει οδηγία ή αρμόδιοι. Το ίδιο θα ισχύει για τις εταιρείες. Αυτή η οδηγία στοχεύει μόνο στα κράτη-μέλη και τις εταιρείες που αρνούνται να κάνουν το οτιδήποτε. Γιατί αυτή θα είναι που σίγουρα θα πρέπει να προσέξουν ότι υπάρχει οδηγία. Και πιστεύω ότι μια οδηγία σε ευρωπαϊκό επίπεδο πραγματικά θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη, και τα κράτη-μέλη όπως η Φιλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και τα υπόλοιπα γιατί οι εταιρείε ε, θα καταλάβουν ότι αν δεν κάνουν αρκετά μέσα στο μοντέλο εκούσιου του κράτους μέλους ε, τότε θα έχουμε περισσότερο δεσμευτικούς κανόνες και εγώ νομίζω ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό κίνητρο για τις εταιρείε ε, για να κάνουν τα όσα πρέπει και να έχουν περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Μάλιστα, ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στο συνάδελφο Γκούναρσον από το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Eh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, πρόσκληση να συμμετάσχουμε στη συνεδρίασή σας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο το να μπορούμε να συζητούμε με τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ανάλυση της κατάστασης δείχνει ότι Με την εισαγωγή νέας νομοθεσία θα μπορέσει να αυξηθεί έως το 2020 σημαντικά το ποσοστό των γυναικών στις ε, μεγάλες επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε ώστε τα ποσοστά να προχωρήσουν, τα αποτελέσματα να βελτιωθούν συνολικά διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε ότι δεν, μπορέσει, θα μπορέσει χωρίς ε, άλλη βοήθεια μέχρι το 2020, ή το 2040 να φτάσει στο 40% ε, συμμετοχή των γυναικών. Αν θέλουμε λοιπόν να επιτύχουμε ένα επίπεδο ισότητας, η ε, προσέγγιση μας θα πρέπει να έχει να κάνει και με τις διαφορές που παρουσιάζονται στην εθνική νομοθεσία, γιατί αυτή μπορεί να οδηγήσει και σε διαφορές στις, στην ανταγωνιστικότητα, στον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Έχουμε να κάνουμε και με διαφορετικές αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει τα κράτη ως προς το θέμα αυτό και έτσι έχουμε κράτη με πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών τα οποία δεν έχουν αναλάβει καμία πρωτοβουλία και θα πρέπει να επιδιώξουν ή να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν τους στόχους αυτούς να τους επιδιώκουν μόνο ε, να τους επιδιώκουν χωρίς να αναλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα. Στην Σουηδία το ποσοστό των γυναικών ήταν 5% στις αρχές του 2000, τώρα έχουμε φτάσει σιγά σιγά στο 20% αλλά πάλι θα πρέπει να ομολογήσουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει μείνει στάσιμο το ποσοστό για να μην πω ότι μειώθηκε ελαφρώς ε, πέρσι και πρόπερσι. Χρειάζεται λοιπόν βεβαίως να προωθήσουμε την αυτορύθμιση σε επίπεδο ε, επιχειρήσω, αλλά όπου χρειάζεται, όπου δεν φέρνει αυτή αποτελέσματα, θα πρέπει και οι κυβερνήσεις να περάσουν στις ε, νομοθετικές ρυθμίσεις. Στην Σουηδία υπάρχει, όπως είπα, η αυτορύθμιση. Δυστυχώς δεν έχει φέρει αποτελέσματα και γι' αυτό θα πρέπει να αναλυφθεί νομοθετική πρωτοβουλία. Ως προς την πρόταση για την οδηγία, ε, χαίρομαι που βλέπω πως έχει πολλά στοιχεία ευελιξίας και επιτρέπει στα κράτη-μέλη να διατυπώνουν τους καρόνες που θεωρούν εκείνα σκοπιμότερους. Ο στόχος του 40% είναι σημαντικός. Είναι σημαντικό επίσης και το χρονοδιάγραμμα που προσδιορίζεται. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο στο οποίο, χρονικό σημείο στο οποίο θα πρέπει να έχει επιτευχθεί πια αυτός ο στόχος. Αλλά βεβαίω θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη κάθε χώρα, χωρί όμω αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να αποδοθεί η ε, μεγάλη ανισότητα στη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια σε εθνικέ ε, ιδιαιτερότητε. Δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε κάτι τέτοιο. Η πρόταση πάντως για παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να πω δεν έχει γίνει δεκτή θετικά από την πλειοψηφία, γιατί εγώ προέρχομαι από το κόμμα της αντιπολίτευσης, από τη μειοψηφία και είμαστε υπέρ της προτάσεως για την οδηγία, αλλά η πλειοψηφία και γενικότερα η κοινωνία των πολιτών στη συζήτηση που έγινε στη Σουηδία τάχθηκε κατά της παρέμβασης επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί επικαλούνται την ε, αρχή της επικουρικότητας. Ωστόσο, και ότι έχουμε αρκετά καλή ε, εκπροσώπηση των γυναικών και παροχές μέρημνα για τα παιδιά, άδειε και ούτω καθεξής, συμμετοχή σε πολύ καλό επίπεδο στο, στην εκπαιδευτική διαδικασία των γυναικών, με ποσοστά καλύτερα από ό,τι αυτά των ανδρών, ε, βλέπουμε ότι αυτό το, αυτή η γυάλινη οροφή δεν έχει διαραγεί ακόμα, δεν έχουν μπορέσει να την περάσουν οι γυναίκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στην Πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών, κυρία Μωρίν Σαρτιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι σήμερα πρέπει πραγματικά να ταρακονηθούμε για το θέμα του προβλήματος των ποσοστώσεων και της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Γιατί γιατί καταρχήν πρόκειται για μία μάχη ισότητας των πολιτών και στην χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων έχουμε εγγράψει αυτή την ισότητα των πολιτών ως μία από τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης. Είναι λοιπόν λογικό να είμαστε όλοι μαζί υπέρ αυτού του στόχου και χαιρετίζω και τις συναδέλφους εισηγήτριες, τις κυρίες Κράτσα και Ρέγνερ, που ανέλαβαν μια τόσο θεμελιώδη έκθεση για αυτή τη νέα οδηγία. Είναι ένας πολύ μεγάλος αγώνας και χαιρετίζω το γεγονός ότι έχουμε μαζί μας πολυάριθμους βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια γιατί όλοι μαζί μόνο θα μπορέσουμε να ελοπίσουμε το στόχο αυτό. Εγώ σας το λέω ειλικρινά. Ήμουν κατά των ποσοστώσεων, ήμουν κατά των ποσοστώσεων του 2000 όταν ε, τις εγκαθίδρυσε η χώρα μου. Γιατί πίστευα ότι οι γυναίκες ε, θα κατάφεραν με τις ικανότητες τους να κατακτήσουν ε, τις θέσεις αυτές. Δέκα χρόνια μετά συνειδητοποίησα ότι είχα κάνει λάθος τα δημόσια χρήματα και τα χρήματα του ιδιωτικού τομέα που επενδύονται στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών για την ε, ισότιμη εκπαίδευση κοριτσιών και αγοριών και επενθυμίζω ότι είπε συνάδελφε προηγουμένω, 60% των πτυχηγών είναι γυναίκες. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε σήμερα ότι αν, έχουμε, αν δεν έχουμε αυτή τη στρατηγική βούληση να ψηφίσουμε για να φτάσουμε στο 40% των γυναικών ε, στα διοικητικά συμβούλια, ποτέ δεν θα τα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Και σας υπενθυμίζω πολύ πρόσφατες αναλύσεις, συγκεκριμένα για την Ιαπωνία, που μας δείχνουν πόσο αυτή η χώρα με τις ε, ιδιαίτερα ματσοπολιτικές που αποκλείουν τις γυναίκες ε, πώς η χώρα αυτή είπα να χωρεί σε διεθνές επίπεδο και σήμερα υποχρεούται να αλλάξει στάση. Ε, ελπίζω ότι εμείς ε, δεν θα φτάσουμε σε τέτοιες ακρότητες. Ήθελα εδώ να υπογραμμίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η οδηγία. Πιστεύω ότι σήμερα οι κατάλογοι των γυναικών που θα μπορούσαν δυνάμει να μπουν στα διοικητικά συμβούλια είναι ένα εργαλείο εντελώς απαραίτητο, Έχουμε πάρα πολλέ ε, γυναίκες που είναι και διαθέσιμε, αλλά πιστεύω ότι και η δημοσίευση των κενών θέσεων στα διοικητικά συμβούλια και των υποψηφιωτήτων ε, είναι κάτι εντελώς ουσιαστικό. Γιατί ξέρουμε ότι πολλές φορές ε, σήμερα έχουμε κάποιες συμφωνίες μεταξύ φίλων, μεταξύ ανδρών. Εγώ δεν είμαι καθόλου κατά των ανδρών, δεν πρέπει να το δείτε έτσι, δεν είναι θέμα φεμινισμού εδώ είναι ένα θέμα ισότητας των πολιτών. Όμως αυτές οι διευθετήσεις μεταξύ φίλων, ε, οι προσλήψεις που γίνονται σε κλειστά κλαμπ, θα πρέπει να λάβουν τέλο. Θα πρέπει η Ευρώπη να βάλει τέλο σε όλα αυτά. Γιατί πίσω από αυτό το πρόβλημα, αν δεν το λάβουμε σοβαρά υπόψη, υπάρχει το πρόβλημα τη σταδιοδρομία των γυναικών που απειλείται. Και βλέπουμε ότι σήμερα οι σταδιοδρομίε των γυναικών ε, δεν εξελίσσονται τόσο όσο οι σταδιοδρομίε των ανδρών. Και θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει και αυτό το πρόβλημα τη σταδιοδρομία των γυναικών, γιατί είναι ένα συνολικό πακέτο το οποίο θα πρέπει να το συνταράξουμε. Ευχαριστώ, Ελιζαμπέτ. Και θα δώσω το λόγο σε μία ακόμη εκπρόσωπο του Συνδικού Κοινοβουλίου, την κυρία Σέντερφελτ. Eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μας απευθύνατε. Είναι ενδιαφέρον ε, να είμαστε εδώ πέρα, να συζητάμε την πρόταση οδηγίας της Κομισιόν. Είμαστε συνάδελφοι από άλλα κοινοβούλια και βεβαίω έχουμε και εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ είμαι μέλος ε, ενός κόμματος που ε, είναι στον κυβερνητικό συνασπισμό της ε, Σουηδίας ε, το μετριοπαθές το λεγόμενο κόμμα μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το ζήτημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να έχουμε ισότητα στα διοικητικά συμβούλια και θεωρούμε πως το γεγονός πως η Κομισιόν έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία είναι κάτι το θετικό. Αλλά Νομίζω πως η πρόταση αυτή δεν ε, συμβάζεται με κάποια εθνικά χαρακτηριστικά. Στην ε, Σουηδία, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι μέτοχοι ε, επηρεάζουν τη σύνθεση του δουσού και τον διορισμό των μελών. Και νομίζω δείχνει αυτό πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα όταν σχηματίζεται ένα διοικητικό συμβούλιο, ε, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και όχι να διορίζεται με βάση το εργατικό δίκαιο. Ε, και είναι υπόλογο το δουσού στους ιδιοκτήτες της εταιρείας, οι οποίοι έχουν τελικά την εξουσία και μπορούν να εξαναγκάσουν τα μέλη του δουσού σε παρέτηση. Οπότε, ο κανονισμός αυτός ε, θα καταλήξει σε μια κατάσταση όπου το αντιμετωπίζουμε το ζήτημα από τη σκοπιά του εργατικού δικαίου, όπου τελικά θα ορίζει ο νόμος την ε, σύνθεση του δουσού και αυτό δεν συμφωνεί με τις Σουηδικές αρχές. Και ε, εγώ και η πλειοψηφία των πολιτικών στην Σουηδία Θεωρούμε πως οι πτυχές αυτές, οι ευρωπαϊκές του ζητήματος δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε χρειάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία ούτε θεωρούμε πως θα αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο. Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι ιδιοκτήτες των εταιριών για να ορίζουν τα μέλη του ΔΣΟΥ είναι νομίζω θέμα του κάθε κράτους μέλους. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κάθε χώρα να βρει τα δικά της μέτρα για το πώς θα αυξηθεί η ισότητα στη βιομηχανία και στα δουσου... Οι εισηγμένες εταιρείε ε, στη Σουηδία έχουν έναν κώδικα ο οποίος αποτελεί τη βάση επιλογής και βεβαίως ε, και στον κανονισμό υπάρχουν κάποιοι κανόνες που μιλάνε για μεγαλύτερη ισότητα των φύλων στα δεσού, αλλά το να αλλάξει η νοοτροπία των ιδιοκτητών των εταιριών είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε με κάποια προγράμματα, προσπαθούμε να επηρεάσουμε για το πώς θα έχουμε περισσότερες γυναίκες. Επιπλέον, η πρόταση ε, έχει αποσταλεί σε επιτροπές ε, στην Σουηδία για διαβούλευση και την απέρριψαν. Ε, ήταν η Σουηδική Ένωση Τραπεζών ε, και η Σουηδική Ακαδημία και οργανώσεις γυναικών και, και τα συνδικάτα επίσης ε, η Συνομοσπονδία των Συνδικάτων ε, έχει θετική άποψη εκτός από ένα συνδικάτο μέλος και επίσης ε, και ο διαμεσολαβητής. Ε, τα μέτρα λοιπόν θεωρούν πως πρέπει να ευθυγραμμιστούν με την κατάσταση που επικρατεί στο κάθε κράτος μέλος, να λάβουν υπόψη της μορφές ιδιοκτησίας και την υπόλοιπη εθνική νομοθεσία. Η νομοθεσία λοιπόν αυτή δεν νομίζω η κατάσταση, με συγχωρείτε, δεν νομίζω πως απαιτεί αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και θα έχει ως αποτέλεσμα παρέμβαση στην, ε, στο πώς διοικούνται οι εταιρείε. Θεωρούμε λοιπόν πως η ισότητα στα διοικητικά συμβούλια είναι σημαντική και στις προτεραιότητας και στη Σουηδία και οπωσδήποτε και σε άλλες χώρες, απλά δεν νομίζω ότι είναι αυτή η σωστή προσέγγιση. Ευχαριστώ κυρία Γκουρμάη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να έχουμε μια τέτοια κοινή συνεδρίαση. ορίζω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και θα ήθελα να γίνεται τέτοια συζήτηση και σε άλλα σημαντικά θέματα με τους συναδέλφους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι βεβαίως πάντα να βλέπω άντρες που ασχολούνται με τα θέματα ισότητας. Και ε, εύχομαι κάθε συνάδελφος να είναι σαν την Ελίζαβεθ ε, ε, από την δεξιά που θεωρούν πως οι γυναίκες ε, είναι ε, η προσθέμενη αξία. Και βέβαια αν, αν έναν άντρα, εκπαιδεύεις μόνο έναν άντρα. Αν εκπαιδεύεις γυναίκες, εκπαιδεύεις γενιές. Και Βεβαίως ε, ακούσαμε τις απόψεις των συναδέλφων για τις ε, ποστός. Είχαμε κάποιες έντονες αντιδράσεις από κράτη-μέλη και τον ε, ιδιωτικό τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να εξηγήσω ποια είναι αυτή η πρόταση και γιατί δεν θα βλάψει τις επιχειρήσεις αλλά αντιθέτως θα φέρει προσθέμενη αξία επιπλέον. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το, το υπάρχον ταλέντο και μην ξεχνάμε πω οι γυναίκες είναι οι περισσότερε από αυτή των πανεπιστημίων, αλλά υποεκπροσωπούνται. Να σα δώσω το παράδειγμα της Ουγγαρία. Οι γυναίκες ε, είναι... Οι γυναίκες έχουν περισσότερα πτυχία από τους άντρες, αλλά δεν ισχύει το ίδιο στα... Αλλά υποεκπροσωπούνται στα δουσού. Οπότε απλά τα, τα πράγματα. Θα έλεγα η συμμεταχείριση όταν γίνεται η επιλογή. Και επίσης πρέπει να επιμείνουμε στις αρχές μας ε, και στο βασικό μας στόχο. Δηλαδή οι γυναίκες και άντρες να έχουν ίσες ευκαιρίες στην πραγματικότητα. Τώρα κατά την άποψή μου η άποψη δεν η πρόταση με συγχωρείτε δεν είναι αρκετά ε, ισχυρή. Ε, το 40% μιλάει για μη εκτελεστικά συμβούλια όπως εποπτικά συμβούλια και δεν είναι εκεί πέρα που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Και μιλάμε και για ευελιξία κτλ. Αντιλαμβάνομαι πως οι κυρώσεις μετά παραμένουν στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, αλλά φοβάμαι πως χωρίς δεσμευτικά μέτρα και κυρώσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο οι οδηγίες αυτές ε, θα, δεν θα έχουν και πολύ νόημα. Χρειάζεται λοιπόν ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριμένα και δεσμευτικά μέτρα, αλλιώς όλα τα άλλα είναι ευσεβής πόθη. Και βεβαίως ε, ε, βλέπουμε το τι προβλέπεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να το δούμε αυτό για τη σωστή ισορροπία. Επιπλέον ανησυχώ για τις προθεσμίες που προβλέπονται για το 2028 για το 30%. Νομίζω πως μπορεί να γυρίσει boomerang και μπορεί να ερμηνευθεί ε, λανθασμένα. Βεβαίως είναι ένα εργαλείο υποσωστώσεις και τελειώνω. Θα ήθελα να πω πως επαφείται σε εμά τώρα να φροντίσουμε η οδηγία αυτή να επιτύχει τον στόχο της, να βελτιώσει την ισότητα και να φτάσουμε τελικά σε ισότητα στο επίπεδο λήψης αποφάσεων. Όπως είπα, είναι όλα αυτά θετικά και για την οικονομία πέρα από την ισότητα και τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Βάγκαπλ από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία που έχω να τοποθετηθώ στην ακρόαση σα για την έκθεση για τη συμμετοχή των γυναικών. Εκπροσωπώ την ε, σοσιαλδημοκρατική ομάδα στο γερμανικό Bundestag, στη Γερμανική Βουλή. Υποστηρίζουμε την πρόταση αυτή όπως την έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερος και την, ε, τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Νομική Επιτροπή και την Επιτροπή των Γυναικών που πιστεύουμε ότι μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση γιατί η κατάσταση όπως έχει τώρα δεν είναι ικανοποιητική, δεν αρκούει δηλαδή τα κράτη-μέλη να δηλώνουν ότι θέλουν να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών. Πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνει αυτή η προσπάθεια και ιδιαίτερα στο χώρο της οικονομίας θα πρέπει να αναδεθούμε σε κοινέ προσπάθειες, να αποδοθούμε σε κοινέ προσπάθειες. θέλουμε λοιπόν συγκεκριμένες θέσεις εμείς στη Γερμανία. Έχουμε συνάψει μία συμφωνία το 2001 ήδη με, την, ε, με το χώρο των επιχειρήσεων ε, για αυτοδέσμευση με αποτέλεσμα τώρα 12 χρόνια μετά, σχεδόν μηδενικό, δεν έχει καθόλου βελτιωθεί χάρη στην εθελοντική αυτή αυτοδέσμευση η παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων και ως εκ τούτου εμείς ως δημοκρατική ομάδα αλλά και η στα κοινικότερα θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να εισαχθούν για ε, δεσμευτικές ε, νομοθεσίες, αλλά δεν έχουμε την πλειοψηφία στο γερμανικό Bundestag γι' αυτό. Ωστόσο υπάρχει το Bundesrat, η Άνω Βουλή, η οποία δεν εκπροσωπείται σήμερα εδώ και η οποία το Δεκέμβριο του 2012 τοποθετήθηκε απερίφραστα υπέρ της ε, υποστήριξης της οδηγίας αυτής και στη Γερμανία με δεσμευτικές ρυθμίσεις. Εάν μου επιτρέπετε θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ σε δύο ζητήματα και να υποστηρίξω τις προτάσεις κυρία Ρέκνερ εκεί όπου αναφερθήκατε στις, ε, στην ιδέα να ζητήσετε πιο ε, αποφασιστική παρέμβαση από αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι δεδομένων ε, των διαφορετικών εταιρικών δικαίων στα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι εύκολο να ε, ε, ερμηνευθεί. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε μια οδηγία που αναφέρεται μόνο σε διοικητικά συμβούλια. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για διοικητικά συμβούλια, αλλά, συμβούλια μη εκτελεστικά μέλη δηλαδή, αλλά για πραγματικά εκτελεστικά όργανα, και αυτό το λέω διότι βλέπουμε ότι στα εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων βλέπουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. 3% είναι μόνο η εκπροσώπηση των γυναικών ενώ είναι 97% οι άντρες. Ε, στις μεγάλες επιχειρήσεις και όταν γνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις, οι πραγματικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο επιχειρήσεων δεν, δεν λαμβάνονται στα εποπτικά συμβούλια αλλά στα... Στα διοικητικά συμβούλια που έχουν εκτελεστικές εξουσίες, ε, προφανώς πρέπει εκεί πέρα να γίνει η παρέμβαση. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε στα εκτελεστικά διοικητικά συμβούλια, ε, στα διοικητικά συμβούλια με εκτελεστικέ αρμοδιότητε, μόνο 3% εκπροσώπηση των γυναικών, 97% είναι οι άντρε. Αυτό δείχνει ότι η δικτύωση μεταξύ των ανδρών είναι τέτοια που ακόμη και όταν οι γυναίκε έχουν πολύ καλή ε, κατάρτιση και δεξιότητε, δεν έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν σε αρότερε θέσει, σε αποφασιστική σημασία θέσει ε, στις επιχειρήσεις. Γι' αυτό σας υποστηρίζουμε και ως προς την πρόταση για τις κυρώσεις, διότι θεωρούμε ότι ε, μπορούμε να έχουμε όσες καλές ε, διακηρύξεις, θέσεις, νομοθετήματα, προτάσεις, αλλά εάν δεν συνοδεύονται αυτά από κυρώσεις δεν φέρουν αποτέλεσμα. Γι' αυτό προκειμένου να βοηθήσουμε να επιτευχθεί συγκεκριμένο αποτέλεσμα στα κράτη-μέλη υποστηρίζουμε την ιδέα για κυρώσεις και ιδιαίτερα την ιδέα την άλλη σας ιδέα, η οποία έχει να κάνει με την υποχρέωση για δημόσια προκήρυξη, γιατί έτσι μπορούμε να, ζητή, να απαιτήσουμε από την ε, επιχείρηση να συμμορφωθεί και να ανοίξει τις, ε, πόρες, τις πόρτες των διοικητικών της ε, συμβουλίων και σε γυναίκες σε εκτελεστικές θέσεις. Ξέρετε ότι στη Γερμανία έχουμε το Σεπτέμβριο εκλογές, θα ανανεωθεί η Βουλή, εγώ ως Δημοκράτης ε, φυσικά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε πολιτική κατεύθυνση στη Γερμανία και ότι έτσι ίσως ανατραπούν και οι ε, τάσεις ε, και οι πλειοψηφίες στην ε, Bundestag προκειμένου να συμφωνήσουμε με μεγαλύτερη πλειοψηφία στην πρόταση αυτή από πλευράς Γερμανίας. Θα δώσω τώρα το λόγο σε άλλο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Λεωτάρ. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβουλία και να τους καλωσορίσω γιατί πραγματικά είναι αναγκαίο να ανταλλάσσουμε απόψεις για το θέμα αυτό. Επιπλέον θα ήθελα να πω πως ε, είμαι υπέρ της ε, ισότητας όλων των φίλων σε όλες τις ε, σφαίρες και στα διοικητικά συμβούλια, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ πέρα. Θα ήθελα Επίσης να πω πως το μέσο των ποστώσεων μπορεί να είναι μια λύση για το θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλα τα επαγγέλματα. Αλλά ε, είναι απλά για να ξεκινήσουμε. Δεν θεωρώ πως θα πρέπει να είναι ένα μόνιμο μέσο. Θεωρώ πως είναι αναγκαίο για να καταπολεμηθεί φτώχεια των γυναικών ε, και των ηλικιωμένων γυναικών. Παρ' όλα αυτά, ε, έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Θεωρώ πως ε, φαίνεται πως η οδηγία δεν αντιλαμβάνεται τη σημερινή κατάσταση, την επισφάλεια των γυναικών ε, στην ε, καθημερινή ζωή σε καιρούς κρίσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η οδηγία αυτή είναι ένα μεγάλο βήμα προς σωστή κατεύθυνση και συνεισφέρει στην μείωση της ανισότητας των φύλων στον τομέα της εργασίας και έτσι θα κλείσει το μισθολογικό χάσμα. Αλλά αυτό γίνεται με έναν τρόπο που δεν είναι ισορροπημένος. Δηλαδή μιλάμε μόνο για διευθυντικές θέσεις και υπάρχει η ψευδέστηση ότι αν έχουμε πολύ περισσότερες γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις θα μειωθούν οι ανισότητες και στις, ε, ε, στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ε, που επιτρέπουν βεβαίως στις γυναίκες να ανέλθουν σε μια τέτοια διευθυντική ε, θέση, αλλά τι γίνεται ταυτόχρονα γίνονται πάρα πολλές οικονομίες και περικοπές και οι γυναίκες ε, χάνουν τις δουλειές τους ή έχουν μόνο προσωρινές δουλειές ή part-time κτλ. Και ε, γίνεται άρα χειρότερη η κατάσταση στον τομέα της ε, ισότητας. Οπότε εάν είναι να γίνουν αυτές οι προτάσεις, πράγματι αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα, ε, εντάξει, παρά το ότι έχουμε εδώ πέρα διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την επικουρικότητα, αν αυτό πρέπει να επιβληθεί από την Ευρώπη, αν πρέπει να γίνει από τα κράτη-μέλη. Θεωρώ πως εάν συμφωνήσουμε κάτι εδώ πέρα, δεν πρέπει να ξεκινήσουμε από την κορυφή, αλλά από τα κατώτερα κλιμάκια. Έτσι θα αγγίξουμε πολύ μεγαλύτερες μάζες γυναικών που θα έχουν πραγματικά την πραγματική δυνατότητα να φτάσουν σε διευθυντικές θέσεις και τότε θα λυθεί το πρόβλημα των φύλων και της ανισότητας στις επιχειρήσεις και η φτώχεια άρα. Επιπλέον, πραγματικά θα ήταν πολύ περίεργο να λέμε πως θέλουμε να μπει ε, ποσόστοση στα κράτη-μέλη, στα δουσού και να μην ε, επιβάλλουμε το 50-50 ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κομισιόν, Κοινοβούλιο, Κεντρική Τράπεζα κτλ. Οπότε εγώ θεωρώ πως πρέπει να έχουμε παντού ισότητα, ναι, αλλά είμαι κάπως δίβουλη όσον αφορά το να μιλάμε για καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία δεν ξεκινάει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μαρτέ, εκπρόσωπο του Ουγγρικού Κοινοβουλίου. Καλημέρα σας, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να εκφράσω την ευχαριστία μου για την ε, σπουδαία αυτή ευκαιρία που μας δίνετε να συμμετάσχουμε στην συνεδρίασή σας και ταυτόχρονα να σας ενημερώσω για τις ε, θέσεις της Ουγγαρίας ως προς την προτινόμενη αυτή οδηγία του Συμβουλίου για την ε, ανατροπή της υποεκπροσώπησης των γυναικών στα ε, διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσει. Σίγουρα και η κυβέρνηση συμφωνεί ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα, για ένα φαινόμενο ε, παγιωμένο, εδρεωμένο, δεν έχουν ε, ε, φέρει προσπάθειες που έχουν αναλυφθεί σε, εθνικό επίπεδο ε, αποτελέσματα και γι' αυτό είμαστε υπέρ μιας προσπάθειας για βελτίωση των ποσοστών αυτών. Αλλά υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι και συνθήκες οι οποίες εξηγούν το φαινόμενο αυτό μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Και ενώ γνωρίζουμε ότι ως προς τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα προσόντα ε, διαφορά δεν εμφανίζεται μεταξύ ανδρών και γυναικών, ε, παραμένει αυτή η απόκληση στην ανάληψη των καθηκόντων που σχετίζεται βέβαια και με την αντίστοιχη ανάληψη των ευθυνών για την διαχείριση της οικογένειας. Και έτσι και δεδομένου ότι και το Σύνταγμα της Ουγγαρίας καταγράφει την αρχή της ισότητας των δύο φύλων και ότι έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες και εκστρατείες της ευαισθητοποίησης στον τομέα αυτών. Θα θέλαμε να υποστηρίξουμε με μακροπρόθεσμα προγράμματα, κοινέ αξιολογήσεις, μελέτες, ανταλλαγή εμπειρίας των στόχων χωρίς όμως να επιβληθούν ε, κυρώσεις. Για τις συστάσεις και τον προσδορισμό των ποσοστώσεων θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι σημαντικά, άλλωστε και οι επιχειρήσεις που είναι συγμένες στο χρηματιστήριο της Βουδαπέστης θεωρούν ότι ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο θα βοηθούσε στην ε, πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή με βάση ε, μια καταγραφή που έγινε το Φεβρουάριο φέτος. Θεωρούν ωστόσο ότι το 40% είναι υπερβολικά φιλόδοξο ποσοστό και σημειώνω ότι από τις 31 εισηγμένες επιχειρήσεις μόνο μία ελέγχεται πλειοψηφικά από το κράτος της Ουγγαρίας. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια τις στατιστικές των, ε, της συμμετοχής των γυναικών να τις ε, ε, παληθεύουμε και να τις συγκρίνουμε γιατί δεν είναι ομοιόμορφες και κλείνοντας θα έλεγα. Ότι ε, και τα συνδικάτα μας θεωρούν ότι δεν μπορούν να επιβληθούν υποχρεωτικές διατάξεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιανακουδάκη, έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν πιστεύω ότι μπορεί κανείς να διαφωνήσει εδώ ότι χρειάζεται περισσότερες γυναίκες να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια, στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, στην πολιτική, σε κάθε εκδήλωση της κοινωνικής ζωής και ότι βέβαια μπορούν να προσφέρουν και ότι προσφέρουν πράγματι όπου συμμετέχουν στο κοινωνικό βίο οι γυναίκες και ότι θα ήταν υποφελή για τι ίδιε επιχειρήσει η παρουσία των τέρων γυναικών στα δικαιωτικά του συμβούλια. Τα μέσα με τα οποία θα υλοποιηθεί λοιπόν ο στόχο, ο οποίο είναι όπω είπα αποδεκτό από όλου, είναι αυτά που ε, διαφέρουν ανάλογα με τη θεώρηση του καθενό. Εγώ σε σχέση με τα όσα ακούσαμε από τη συζήτηση αυτή, ε, ανησυχώ λίγο γιατί νομίζω ότι έχει παρεκτραπεί η συζήτηση και δεν αφορά μόνο την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων, είναι μόνο σαν να ε, επιβεβαιώνουμε ένα κατάλογο προϋποθέσεων για τις επιχειρήσεις συγμένες. Πολύ καλά, αλλά οι άλλες επιχειρήσεις, φερειπίν μεγάλες εταιρείες δικηγόρων, μεγάλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείε ε, παροχής ε, συμβουλών οικονομικών ή λογιστικού ελέγχου, γιατί δεν τις περιλαμβάνουμε αυτές και τι είδους δομές είναι αυτές που επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό να παρέμβει στι εθνικέ εθνικά, ε, στις εθνικές νομοθεσίες. Έτσι λοιπόν η εθελοντική προσέγγιση φαίνεται για μένα ως η πιο αποτελεσματική μακροπρόθεσμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε την έκθεση Ντένις η οποία δίνει κάποιες πολύ θετικέ ε, εκτιμήσεις. Παρουσιάζεται δηλαδή κατά 15% από το 12% συγγνώμη, στο 17% και μισό της εκατό αύξηση της παρουσίας των γυναικών χάρη στην εθελοντική προσέγγιση που είχαμε. Αυτό το καταγράφει τελευταία έκθεση μέσα σε ένα χρόνο και άρα μπορούμε να στηριχθούμε σε αυτήν. Οι ιδέες για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, επί παραδείγματι, πάνω στις οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη, η αμοιβαία ενθάρρυνση ε, από το ένα κράτος στο άλλο για να κάνουν μια περισσότερη προσπάθεια. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιβάλλουμε όμως νομοθεσία και κυρώσεις, γιατί σε ένα θέμα το οποίο είναι τόσο διαφορετική, παρουσιάζει τόσο διαφορετική εικόνα σε κάθε κράτος μέλος, οι ανάγκες των κοινωνιών αλλά και των, και των εταιριών είναι τόσο διαφορετικές, που εάν ε, επιμείνουμε το μόνο που θα μπορέσουμε να κάνουμε θα είναι να πέσουμε στην παγίδα που έπεσε η Νορβηγία, δηλαδή να κατασκευάζουμε γυναίκες ε, συμβολικής ε, ε, θέσης, γυναίκες που θα παρουσιάζονται ως τρόπεα, θα έχουν μη εκτελεστικές αρμοδιότητες, όσες και να είναι αυτές οι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια δεν θα έχουν καμία αρμοδιότητα και θα είναι μόνο για το Θεαθήνε. Αυτό, αυτό ήταν τελικά η ιστορία στην Νορβηγία και δεν αυξήθηκε καθόλου η παρουσία γυναικών με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Δεν ξέρω, σε αυτό που είπε η φίλη κυρία Λεωτάρ, ε, αν μπορούμε κάπως να ανοίξουμε το δρόμο για τις γυναίκες, να τις βοηθήσουμε να δραστηριοποιηθούν επιστροφές στις επιχειρήσεις και έτσι να φτάσουν στα υψηλότερα κλιμάκια. Πολλά έχουμε να κάνουμε, πολλά έχουμε να δεχθούμε ένας από τον άλλον και σε αυτό στηρίζομαι και εγώ για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα στο λόγο στο συνάδελφο Ρικάρδο Τρίγες από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να μιλήσω πορτογαλικά, την μπορώ. Μάλιστα, καλημέρα σας, ευχαριστώ. Καταρχήν ε, θέλω να χαιρετήσω την πρόεδρο αυτής της Επιτροπής, την Αντίτα Στρέλα, και να πω ότι σήμερα σε αυτή την Επιτροπή έχουμε ένα Προεδρείο που αποκαλείται αποκλειστικά από γυναίκες και το χαιρετίζω αυτό. Έτσι λοιπόν ε, το θέμα ε, που συζητάμε εδώ μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι η κατάσταση στην Πορτογαλία. Δεν διαφέρει πάρα πολύ από αυτά που ισχύουν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα δημοκρατικά κράτη και τα κράτη δικαίου έχουν το σύνταγμά του όπου η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί δικαίωμα και όλοι ξέρουμε ότι αυτό το αυτή η επιθυμία δεν έχει καλυφθεί από προδραστικά μέτρα, δεν υπήρχε ούτε στο πρωτοκολλικό καθεστώς ποσοστώσεις, παρά μέχρι πριν λίγα χρόνια. Και Όλοι ξέραμε ότι επιθυμούσαμε να υπάρχει συμμετοχή των γυναικών, όμως στην πράξη είδαμε ότι όταν δεν υπάρχει νομοθεσία ισότητας, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στους πολιτικούς θεσμούς. Το ίδιο συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις δηλαδή η έλλειψη ενός προδραστικού μέτρου στις επιχειρήσεις, στην ιδιωτική οικονομία ε, που να αφορά την εκπροσώπηση των ε, γυναικών ε, στα διοικητικά συμβούλια σημαίνει ότι είναι πολύ χαμηλότερη η εκπροσώπηση τους. Έτσι λοιπόν αυτό μας οδηγεί να σκεφτούμε αν θα πρέπει να λάβουμε ένα δεσμευτικό μέτρο ή όχι σε όλα τα κράτη-μέλη. Εγώ νομίζω ότι και στην Πορτογαλία που αυτό το μέτρο δεν είναι κάτι που γίνεται αποδεκτό χωρίς αντιρρήσεις. Ε, παρόλα αυτά είδαμε και την ε, εποχή του κυβερνητικού κόμματος ε, ε, από το θέμα αυτό όμως οι σοσιαλιστές υπερψήφισαν έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι προτείνουμε ένα ριζοσπαστικό μέτρο για τα κρατημέλη. Τελικά όχι όμως, η πρόταση αυτή είναι πάρα πολύ μετριοπαθής, ντροπαλή θα έλεγα για να πετύχει τους στόχους που θέλει. Έτσι λοιπόν ε, μιλάμε εδώ για μη εκτελεστικές διοικητικές θέσεις και μιλάμε για ορισμένα διοικητικά συμβούλια. Δηλαδή όταν μιλάμε για θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών. Από την άλλη, δεν, ε, εδώ δεν μιλάμε για όλες τις επιχειρήσεις, μιλάμε για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και η πρόταση στοχεύει στο να καλύψει μία περίοδο μέχρι το 18-2020 καλύπτει μια συγκεκριμένη περίοδο δηλαδή. Έτσι λοιπόν εδώ τι θέλουμε να έχουμε. Ε, κάποια μέτρα να εθετηθούν κάποια μέτρα που μας φαίνονται προδραστικά και δίχως αυτά τα μέτρα δεν θα είναι δυνατόν να πετύχουμε την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Όπως σας είπα, Υπάρχουν όλες αυτές οι προθέσεις, ε, θεωρητικά όμως στην πράξη έχουμε διότι ότι όταν δεν λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα υπάρχουν και στην Πορτογαλία συστάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που λέει ότι στα διοικητικά συμβούλια θα πρέπει να συμμετέχουν ε, και οι γυναίκες. Όμως ε, βλέπουμε ότι οι συστάσεις αυτές στην πράξη δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα που επιθυμούμε και πρόκειται για ένα μέτρο που σέβεται την αρχή της επικουρικότητας και τα κριτήρια που έχει θέσει ήδη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν δίνουμε επομένως κανένα προνόμιο στις γυναίκες γιατί εδώ μιλάμε για ισότητα των προσόντων και όταν μιλάμε για ισότητα προσόντων, δεν μιλάμε για αυτόματο διορισμό χωρίς να ισχύει κανένα άλλο κριτήριο. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και όταν και ένας άνδρας και μια γυναίκα έχουν ίσα προσόντα, πέραν αυτού υπάρχουν και κριτήρια που δεν είναι αυτόματα και που διέπουν ε, τη διαδικασία της επιλογής. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογική η πρόταση αυτή και που η Πορτογαλία και εγώ πολύ συγκεκριμένα, καθώς είμαι από το κόμμα της ε, αντιπολίτευσης, ε, θα την υποστηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ρικάρντο, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Κοκμέρη τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Mm. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την παράθεση της κυρίας Ρέντινγκ. Είπε ότι πιστεύει ότι οι συναισθηματικές συζητήσεις που έχουν προκαλέσει, που έχουν προκληθεί από την πρόταση της οδηγίας, δεν είναι λόγο του πεδίου εφαρμογής οδηγίας, γιατί ακούσαμε ότι είναι περιορισμένος και ο αριθμό των εταιριών που θα έπρεπε να συμμορφωθούν με την οδηγία περίπου 5.000. Δεν αφορά λοιπόν περισσότερο το πεδίο εφαρμογή, αλλά όλοι ξαφνικά έχουν μία γνώμη υπέρ κατά των ποσοστώσεων. Και είπε ότι δεν τη αρέσουν οι ποσοστώσει, αλλά τη αρέσει το τι κάνουν οι ποσοστώσει. Και βλέπω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ευρία πλειοψηφία υπέρ των ποσοστώσεων και πράγματι αναφέρθηκαν σε αυτό και συνάδελφοι πολλέ φορέ. Έχουμε ζητήσει από την Κομισιόν μέσω ονομαστική ψηφορία να παρουσιάσει μια πρόταση και ε, το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πήγε πολύ μακρύτερα από αυτά που βλέπουμε σήμερα επιτάπητος. Και επίσης βλέπουμε ότι η Επιτροπή των Περιφερειών αλλά και η Οικονομική και η Κοινωνική Επιτροπή ε, και ήδη έχουν γνωμοδοτήσει σχετικά με την πρόταση αυτή και οι δύο επιτροπές αυτές είναι υπέρ. Επομένως, από τους συμβουλευτικούς ε, θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε ότι υπάρχουν θετικές στάσεις κυρία Ρέγνερ και κυρία Κράτσα. Εκτιμώ πάρα πολύ τη σημαντική σας δουλειά για αυτήν την οδηγία. Ήδη αναφέρατε πάρα πολλά από τα σημεία που θέλω να θίξω κι εγώ και μπορώ να πω ότι οι περισσότεροι από τους ελευθέρους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν με όσα υπόθηκαν. Πέρα από τη νομική βάση που προφανώς αποτελεί τη βάση της εργασίας μας, Νομίζω ότι από τη σκοπιά των φιλελευθέρων ε, θα μπορούσε κάποιος να θέσει ξανά το πολιτικό ζήτημα του τι κάνουμε ως νομοθέτες ε, αν ε, δεν υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός, αν δεν είναι δυνατός. Και βλέπουμε ότι και σε άλλους τομείς που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, οι νομοθέτες ε, παρέχουν ένα πλαίσιο για να αποφύγουμε τα λιγοπόλια, παραδείγματο χάρη, να αποφύγουμε τα μονοπόλια, γιατί πιστεύουν οι νομοθέτε στην καινοτομία και ότι οι καλύτερε υπηρεσίε για του καταναλωτέ επιτυχάνονται όταν λειτουργεί ο ανταγωνισμό. Και εγώ νομίζω ότι γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο και σε αυτόν τον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, αν μπορώ να το πω έτσι. Και να ολοκληρώσω λέγοντας ε, ότι από τη χώρα που ξέρω εγώ καλύτερα μπορούμε να περιμένουμε αλλαγές το Σεπτέμβριο και ακόμη και αν το SPD συνεχίζει να έχει χαμηλές προοπτικές να είναι στην κυβέρνηση θα είναι πλειοψηφία στην ε, Κάτω Βουλή, γιατί η ΣΕΝΤΕΟΥ έχει ανακοινώσει ότι ένα από τα σχέδιά του για την επόμενη νομοθετική περίοδο είναι να παρουσιάσει νομικά δεσμευτικέ ποσοστώσει για τη Γερμανία και το SPD και η Πράσινη είναι ήδη υπέρ. Έτσι λοιπόν ε, στην Λιθουανική Προεδρία θα πρέπει να επιμείνουμε. Θα έχουμε διαφορετικές πλειοψηφίες από αυτές που βλέπουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Μασίπιντάλγο από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Στρέλα. Εγώ λυπάμαι που εδώ σήμερα δεν υπάρχει εκπροσώπηση από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Συγγνώμη, κύριε Λούλινγκ. Εγώ είμαι κουτσός και δεν ε, ε μπορώ να χρησιμοποιήσω και τη χέρι μου πρέπει, αλλά έχω πολύ δυνατή φωνή και θέλω να τη χρησιμοποιώ εδώ στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, επομένως, ε, στην Ισπανία αυτό το θέμα ε, είναι σημαντικό και σε πολύ μεγάλο βαθμό είμαστε στην πρωτοπορία για τον αγώνα, για τη μάχη, για την ισότητα μεταξύ των φίλων. κάτι στο οποίο στοχεύει αυτή η νομοθεσία. Υποστηρίζω την κυρία Κράτσα, υποστηρίζω και την κυρία Ρέγκλερ, είμαι μέλος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και όπως είπε και πριν η πρόσωπος των ελευθερών η νομική βάση σήμερα πρέπει να εγκριθεί στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αύριο. Γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί δισταγμοί, υπερβολικοί δισταγμοί από ε, από τη σκοπιά ε, αυτού που λέγαμε πριν ότι το φάντασμα που διατρέχει τον κόσμο είναι ε, ο ματσισμός και Επομένως, δεν παραμένει καμία αμφιβολία πως ε, εξακολουθούν να υπάρχουν επικίνδυνες απόψεις ε, όσων αντιτίθεται σε αυτήν την νομοθεσία. Όμως ε, θέλω να αναφερθώ και σε κάτι ακόμη, όσο λέγονται για τον αγώνα για την ισότητα των δύο φύλων και όσα είπαν κάποιοι για μια επιχείρηση που δεν είχε καμία εκπροσώπηση από το γυναικείο φύλλο. αυτή ε, πραγματικά έδιναν μία πάρα πολύ άσχημη εικόνα προς τα έξω. Έτσι λοιπόν θα πρέπει οι πολίτες να θεωρούν ότι όσοι δεν πληρούν το πνεύμα αυτής της οδηγίας είναι πραγματικά αξιοθρύνητοι. Και αυτό το θέμα της εκπροσώπησης, της ισότητας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην Ευρώπη. Εμείς δίναμε το παράδειγμα, είμαστε παραδειγματικοί σε αυτά, αλλά θα πρέπει να είμαστε παραδειγματικοί και στο σεβασμό της ισότητας των δύο φύλων. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη ισότητα. Πρέπει να μας δίνει το πνεύμα της ισότητας, γιατί όχι μόνο θα το πετύχουμε για την Ευρώπη, αλλά το παράδειγμα θα το δώσουμε σε ολοκλήρω τον κόσμο. Γιατί έχουμε πολλά μέρη στον κόσμο όπου φυσικά η κατάσταση των γυναικών είναι πάρα πολύ χειρότερη και άλλοι πολιτισμοί πρέπει να δουν τα βήματα που κάνουμε εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα βήματα που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να είναι παραδειγματικά και πρέπει να κερδίσουμε αυτή τη μάχη γιατί είναι παγκόσμια, όχι απλώς ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αντώνιο. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Χάνιμπολ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και καλώ ορίζω τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είναι σε μεγάλο βαθμό ενθαρρυντικό το ότι συμφωνούμε επί της αρχής, αλλά από την άλλη είναι και εύκολο να συμφωνούμε επί της αρχής της ισότητας των φύλων και τη ισότητα εν γέννη. Πιο δύσκολο είναι από την άλλη να βρούμε έναν τρόπο την ισότητα αυτή να την υλοποιήσουμε στην πράξη, ώστε να επιτευχθεί πράγματι. Και οφείλω να πω ότι κάποιες από τις απαντήσεις που ακούσαμε εδώ ήταν απογοητευτικές, αν και κάποιες άλλες ήταν πολύ καλές. Από τα Εθνικά Κοινοβούλια προκύπτει ξεκάθαρα, πιστεύω, ότι τα εθελοντικά συστήματα, όσοι και αν είναι η αξία που τους αναγνωρίζεται, δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, επί παραδείγματι, έχουμε 17% γυναίκες στις επιχειρήσεις του Φούτσι 100. Πολύ λίγο. Και όσο καλό και είναι το 17, εμείς ήταν 40%, όχι 50%. Επίσης, λοιπόν, θα ήθελα να πω για εκείνους τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και τις πολιτικές ομάδες ή κόμματα που δεν συμφωνούν με τις ποσοστώσεις. Θα ήθελα λοιπόν να τους πω ότι η νομοθεσία αυτή έχει συνταχθεί με ιδιαίτερη προσοχή και μέρημνα να επιτρέπεται στις χώρες που έχουν ήδη υφιστάμενες θελοντικές συμφωνίες να τις διατηρήσουν εφόσον μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μπορούν να επιτύχουν τις ε, Η κυρία Κορνέλης τον το νωρίτερα που είναι και η συντάκτρια, αλλά δεν το προσέξατε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν ε, ε, που υπάρχουν οι εθελοντικές δεσμεύσεις, εάν φέρουν αποτέλεσμα μέχρι το 2017, όπως φαίνεται θα τα καταφέρουμε, δεν θα χρειαστεί να επιβληθούν τα υποχρεωτικά μέτρα. Γι' αυτό λοιπόν καλό το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, την Ουγγαρία και όλες τις άλλες χώρες που δεν θέλουν την εισαγωγή ε, υποχρεωστικών ποσοστώσεων και την κυρία Γιαννακουδάκη από την ομάδα συντηρητικών μεταρρυθμιστών να δεχθούν το επιχείρημα αυτό ότι χρειάζονται ως ουσιώδη στοιχείο της νομοθεσίας οι ποσοστώσεις και να το δεχθούν συμβιβαστικά γιατί και εμείς από την Επιτροπή των Γυναικών αλλά και από την Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων που είμαι και αναπληρωματικό μέλος θέλουμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Θέλουμε εν τέλει να Υπάρχουν γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια και πιστεύουμε ότι αυτή η νομοθεσία θα μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε το στόχο αυτό, ενώ ταυτόχρονα δεν αποκλείονται άλλες λύσεις που ενδεχομένως έχουν ε, προτιμήσει κάποιοι άλλοι και θα μπορέσουν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις ε, στην επιλογή ε, γυναικών με κατάλληλες δεξιότητες και προσόντα. Βεβαίως και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε να παίρνουν περισσότερες δεξιότητες και κατάρτιση οι γυναίκες, πως αυτό όμως να σημαίνει ότι αποκλείεται και η αξιοποίηση των ποσοστώσεων. Είναι πολύ καλό το νομοθέτημα λοιπόν. Οι χώρες οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει μια πορεία με θελοντική δέσμευση μπορούν να την διατηρήσουν. Κάποιες άλλες όμως θα υποχρεωθούν να φέρουν πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα ως προς την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβουλία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Νίμπλερ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ θερμά ε, τους συναδέλφους, τις συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια που ήρθαν σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συζητήσουν μαζί μας και να ανταλλάξουν απόψεις για το σημαντικό αυτό θέμα. Ε, σέβομαι φυσικά τις διαφοροποιημένες θέσεις που εκφράζονται. Ο στόχος είναι κοινός. Το ζήτημα είναι πώς θα τον επιτύχουμε. Και αυτό είναι και ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, εξασφαλίσει περισσότερε ηγετικέ θέσει για τι γυναίκε, περισσότερη εκπροσώπηση των γυναικών στι ηγετικέ θέσει επιχειρήσει. Άκουσα λοιπόν τα επιχειρήματα. Όσον αφορά τη δική μου πατρίδα, επιτρέψτε μου μία παρατήρηση προ τη συνάδελφο από την Bundestag. Χαίρομαι που είστε εδώ. Καταρχά, αλλά θα ήθελα για λόγου τάξη κιόλα να υπενθυμίσω, γιατί είπατε ότι το S5, οι SND, ε, σοσιαλδημοκράτε, ε, είναι θετική στην ε, θέση αυτή, αλλά στην πρόταση αυτή, αλλά θα σας υπενθυμίσω ότι μέχρι το 2005 που είχατε 7 χρόνια τη διακυβέρνηση της χώρας δεν κάνατε τίποτα για να εισαγάγετε ε, υποχρεωτικέ υποχρεωτικές για την εκπροσώπηση των γυναικών. Δεν είναι τίποτα. Τώρα χάρη, ευτυχώς ε, τώρα πια έχουμε μια πολύ ε, διαφορετική θέση και ανεξαρτήτως της έκβασης των εκλογών θα έχουμε θετικές, ε, υποχρεωτικές μάλλον ποσοστώσεις από το φθινόπωρο και μετά. Ε, ήταν η θέση της Επιτροπής όπως εκφράζεται πιστεύω θετική, ήταν μετριοπαθής, μπορούν να την υποστηρίξουν φανταζόμαι και τα κράτη-μέλη. Η συγγήτρια κυρία Ρέγνερ από την Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων μας επεσήμανε ότι αύριο θα ψηφιστεί η νομική βάση της προτάσεως και ομολογώ ότι έχω κάποιες επιφυλάξεις με την έννοια ότι και είμαι πολιτική εκπρόσωπος του κόμματός μου και είμαι υπέρ της προτάσεως επ' αυτή την έννοια, αλλά ως νομικός αισθάνομαι μια δυστημία γιατί δεν είμαι βεβαία ότι μπορεί το 157.3 να ερμηνευθεί κατά αυτόν τον τρόπο απαραίτητα. Και δεν είμαι βεβαία ότι έχει αρμοδιότητες νομοθετικές η Ένωση στην υπόθεση αυτή. Θα δούμε όμως με την έκβαση της ψηφοφορία ε, ίσως τελικά να υποστηρίξει τη νομική αυτή βάση πλειοψηφία των συναδέλφων στην Νομική Επιτροπή. Αλλά πάντως από νομική άποψη για μένα υπάρχουν κάποια σημαντικά ερωτηματικά. Θα γίνει βέβαια η συζήτηση, θα συνεχιστεί η συζήτηση. Χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα εδώ να κάνουμε μια εντατική συζήτηση, να διαμορφώσουμε άποψη, να παρακολουθήσουμε ποια είναι η κατάσταση και στα κράτη-μέλη και περιμένω βέβαια να δω την έκθεση στην, ε, με την πρόταση εκθέσεως για να καταθέσουμε και εμείς τροπολογίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λίχτενμπεργκερ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς και εγώ το θέμα αυτό ήθελα να θίξω την νομική βάση που είναι πράγματι ένα θέμα καυτό γιατί είναι θέμα αρχών. Εγώ ήμουν μέλος Ευρωπαϊκής, μέλος Ευρωπαϊκής Συνέλευσης και ήταν πάρα πολύ σημαντικό να λειτουργήσει και ο κατάλογος των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εδώ όμως που έχουμε να λάβουμε μία απόφαση μεταξύ επικουρικότητας και επιχειρημάτων που λύνονται μόνο τους, αρκεί να περιμένει κανείς γύρω στα χιλιά χρόνια περίπου, αλλά θα γίνει κάποτε. Πρέπει να σκεφτούμε και ε, τη νομική βάση Ε, κοιτάξτε, ε, όταν μιλάμε για νομική βάση και οι γνωμοδοτήσεις δεν είναι πάντα αντικειμενικές. Ε, εγώ είμαι πεπισμένη πως στέκει η νομική βάση. Η ιδέα αντίρρηση περί επικουρικότητα στο πλαίσιο αυτό έχει ένα πρόβλημα, γίνει ένα πρόβλημα, γιατί η ποσόστοση δεν, δεν είναι το πρώτο εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί και λέμε τώρα θα μπει ποσόστοση παντού, αλλά υπάρχει μία περίοδος ε, κατά την οποία έχουν τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να ορίσουν κάποιες αρχές ε, σε διάφορους τομείς και να τις επιβάλλουν. Ε, υπενθυμίζω και άλλα θέματα. Θελοντική δέσμευση της βιομηχανίας σε πολλούς κλάδους που δεν οδήγησε στην επίτευξη των στόχων. Οπότε με την εθελοντική αυτή δέσμευση δεν είχαμε αύξηση της συμμετοχής των γυναικών ούτε κατά 1%. Ε, και τώρα πάμε στο επόμενο βήμα. Επικουρικότητα. Η επικουρικότητα κατά την άποψή μου δεν είναι το τελειωτικό επιχείρημα εδώ πέρα. Δηλαδή ότι δεν μας αρέσει λέμε επικουρικότητα. Και δεν πρέπει να ρυθμίσουμε τα πράγματα ευρωπαϊκά. Θεωρώ πως ε, από τις ευρωπαϊκές συνθήκες προκύπτει κάλλιστα η δυνατότητα αυτή και θεωρώ πως η ποσόστοση αυτή τη στιγμή είναι ένα αποφασιστικό βήμα. Δεν προέκυψε ε, έτσι από το πουθενά πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Περιμέναμε την αυτορύθμιση, δεν έγινε. Τώρα έχουμε την επιλογή είτε να περιμένουμε άλλα 200 χρόνια ή έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, θεωρώ πως επί της ουσίας συμφωνούμε. Έτσι. Ε, η συμμετοχή των γυναικών στα δουσού δεν είναι μόνο θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά θα έχει και θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή αυτά τα, αυτές οι κλειστές αντρικές λέσχες. Δεν νομίζω να τα πήγαν και τόσο καλά στο παρελθόν, δεν στέκει και οικονομικά. Άρα το επόμενο βήμα είναι νομίζω ενδιαφέρον. Γι' αυτό χαίρομαι για αυτή τη συζήτηση και με τους εθνικούς βουλευτές και με τις εμπειρίες που ανταλλάξαμε σήμερα ε, να προχωρήσει νομίζω η συζήτηση και στο εθνικό πλαίσιο. Θα ληφθεί υπόψη η επικουρικότητα. Στην πρόταση ε, αναφέρεται ωραιότατα και θεωρώ πως θα ήταν ωραίο στο τέλος αυτής της θητείας να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα ε, στον τομέα της πολιτικής των γυναικών. Και απευθύνω έκκληση σε αυτούς που πιστεύουν στην επικουρικότητα, σκεφτείτε πως καμιά φορά και άλλες πρωτοβουλίες που δεν ανήκουν στην επικουρικότητα είναι θετικές. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στους κυρίους Λούλιν και Κλέβεν. Αλλά είστε πάρα πολύ σύντομε γιατί θα πρέπει να δώσω το λόγο και στις συνσηγήτριες. Ναι, θα είμαι πολύ σύντομη κυρία Πρόεδρε. Θέλω να πω καταρχά ότι ή τι άλλο πρέπει να επενέσουμε την Επιτροπή γιατί τάραξε τα νερά ως προς την εκπροσώπηση των γυναικών στα ε, όργανα λήψη αποφάσεων σε κάθε τομέα, αλλά αυτή η, απόφαση, αυτή πρόταση μάλλον αφορά μόνο τα όργανα λήψη αποφάσεων σε επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Εφόσον εφαρμοστεί, θα εξασφαλίσουμε το πολύ πολύ καμιά δεκαριά γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια ή στα εποπτικά συμβούλια των επιχειρήσεων ε, των εισηγμένων στις επιχειρήσεις. Δεν θέλω να πω δε ότι, όπως έχει ήδη επισημανθεί, είναι πολύ διαφορετικό το εταιρικό δίκαιο στα κράτη-μέλη. Στη Γερμανία υπάρχει το Aufsichtsrat, υποπτικό συμβούλιο, ενώ το Λουξεμβούργο έχει δομές αντίστοιχες με αυτές της Γαλλίας, με διοικητικό συμβούλιο. Και εδώ οι διαφορές είναι τεράστιες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε μια ευρωπαϊκή οδηγία που θα χειρίζεται τα θέματα που αφορούν τα δύο, τους δύο αυτούς τύπους συμβουλίων, ε, οργάνων, λήψη αποφάσεων με τον ίδιο τρόπο. Για δε τη νομική βάση δεν με καν βεβαία ότι είναι πρόσφορη για τη θέσπιση οδηγίας για τα διοικητικά συμβούλια αποκλειστικά επιχειρήσεων εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Ε, σημειώθηκε ότι υπάρχει μια πλειοψηφία που είστε υπέρ των ποσοστώσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ θα ήθελα να πω το εξή, ότι ο χειρότερος εχθρός της πολιτικής που επιδιώκει πραγματική εκπροσώπηση, καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών, θα είναι όλοι αυτές και αυτοί, όλες και όλοι αυτές και αυτοί που υπερβάλλουν στις διεκδικήσεις τους. Και σημειώνω, ύστερα από τα όσα άκουσα, και από εκείνους ή εκείνες που ζητούν ακόμη και δημόσια προκήρυξη χειρευουσών θέσεων και ανοιχτές διαδικασίες για πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Είναι υπερβολικό αυτό. Έτσι λοιπόν εγώ αυτό ε, που φοβάμαι περισσότερο δεν είναι τα ερωτήματα που ενδεχομένως διατυπώνει κάποιος από εμά, αλλά φοβάμαι περισσότερο αυτούς και αυτές μεταξύ μας που συχνά και πολύ συχνά δυστυχώς στη δική μας περίπτωση όπως στην Επιτροπή των Γυναικών διατυπώνουν ακραίες υπερβολικές διεκδικήσεις που καθιστούν γελίο το Κοινοβούλιο και που δυστυχώς ενισχύουν τις θέσεις στο Συμβούλιο εκείνων που δεν θέλουν να ακούσουν να γίνεται λόγος για τέτοιου είδους ισότιμη εκπροσώπηση και τελικά μόνο κακό κάνουν σε αυτόν τον αγώνα και σε αυτόν τον στόχο. Αρκετά είπα, αλλά πρέπει να πω ότι φοβούμε πράγματι ότι και με βάση τα όσα έχω ακούσει μέχρι τώρα ότι οι θέσεις μας όπως εκφράζονται δεν θα ληφθούν σοβαρά υπόψη από το Συμβούλιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κλέβα, παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Είμαι σύντομη, θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Σήμερα μιλάμε για την διαφορά την ενοιολογική μεταξύ εθελοντικών και υποχρεωτικών μέτρων. Εγώ πιστεύω στις ποσοστώσεις γιατί έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές. Θεωρώ πως θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες στην οικονομία, στις εταιρείες. Ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα στην Επιτροπή Οικονομικών και θα ήθελα να επισημάνω την πολύ σημαντική πτυχή που δεν αναφέρθηκε. Υπάρχουν μελέτες ε, που ε, ασχολούνται με τις ποσοστώσεις εταιρείε, οι οποίες έχουν καταδείξει πως είναι υποφελείς οι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Η λειτουργία εταιριών με μικτές ομάδες, με μεγάλη εκπροσώπηση γυναικών στο έχει βελτιωθεί. Τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα κάθε χρόνο που περνούσε. Και είναι ενδιαφέρον όταν μιλάμε για εταιρείε. Ο κόσμος δεν έχει προβλήματα με την ποσοστοσή, δεν έχει προβλήματα με τις γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις, σε αντίθεση με την πολιτική παραδείγματος χάρη. Προσωπικά θεωρώ πως δεν πάμε αρκετά μακριά πρέπει να ζητήσουμε το 50%. Δεν ξέρω γιατί σταματήσαμε στο 40%. Εάν στο κοινοβούλιο, όταν το συζητάμε δημόσια δηλαδή, εάν μειώνουμε εμείς από μόνες μας ε, τις φιλοδοξίες μας, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Πρέπει να κάνουμε και περισσότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν να δώσω το λόγο στις συνεισηγήτριες, θα ήθελα για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια για την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους εδώ στη συζήτηση. Συνήσφεραν πάρα πολύ στον εμπλουτισμό της συζήτησης, μας έδωσαν διάφορες οπτικές. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η συζήτηση, ιδιαίτερα επικοδομητική και επίσης ήταν ε, και χρήσιμη για τις εισηγήτριες που προφανώς ε, θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματα. Και να επενθυμίσω πως το χρονοδιάγραμμα για αυτή την έκθεση θα είναι το εξής τον Ιούλιο είτε στις 8, είτε στις 9, είτε στις 10. Θα έχουμε παρουσίαση της έκθεσης. Κατόπιν θα κατατεθούν τροπολογίες μέχρι τις 29 Αυγούστου, στις 5 το απόγευμα. Η συζήτηση των τροπολογιών θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου και η ψηφοφορία στις Επιτροπής Γιούρι και ΦΑΜ στις 14 Οκτωβρίου. Λαχθέντων αυτών, να ζητήσω λίγο παραπάνω χρόνο από τους διερμηνείς και τους ευχαριστώ για τη δουλειά τους γιατί μας βοηθούν να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Ευχαριστώ λοιπόν τους διερμηνείς να δώσω στην κυρία Κράτσα το λόγο για τα τελικά συμπεράσματα Θα σας ζητήσω να είστε πολύ σύντομοι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για αυτή τη συνάντηση και τη συζήτηση που έγινε σήμερα με τους με τους άνδρες και γυναίκες εκπροσώπους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και να ευχαριστήσω επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρουσίασε τις κρίσιμες πτυχές της ε, οδηγίας καθώς και την Προεδρία, την ε, Ιρλανδική και την Λιθουανική και περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον τις προτάσεις που μας ε, υποσχέθηκαν. Επίσης, παρόλο που δεν πήραν το λόγο, πρέπει να ευχαριστήσουμε και τα δύο συμβουλευτικά μας όργανα, την Επιτροπή Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για την προσοχή με την οποία ασχολήθηκαν και τις ε, ε, γνώμες τις οποίες μας εξέδωσαν. Ε, συμπερασματικά διαπιστώσω, διαπίστωσα και πιστεύω το μοιράζομαι μαζί σας ότι υπάρχει ακόμη μια διστακτικότητα τόσο στην κοινή γνώμη και στα ε, διάφορα πολιτικά κόμματα ε, σε σχέση με την οδηγία, το στόχο που υπηρετεί και τη μέθοδο που θα τον υπηρετήσει. Ε, πιστεύω όμως ότι η συζήτηση που κάναμε σήμερα ε, θα καταλήξει σε κάποια σύγκληση. γιατί διευκρινίστηκαν κάποια θέματα πάρα πολύ βασικά, κυρίως για τους συναδέλφους που διστάζουν ακόμη. Ε, παραδείγματος χάρη, ε, το, το, επιχείρημα ότι δεν έχουμε το ίδιο εταιρικό δίκαιο στις διάφορες ε, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που το έχουμε και εμείς αναφέρει. Η οδηγία όμως δεν ενοχλεί, το πεδίο οδηγίας δεν ενοχλεί τα εταιρικά ε, δίκαια, διότι εφαρμόζεται στο όργανο το μοναδικό ή στα όργανα που έχουν μη εκτελεστικά μέλη. Οπότε αυτό πιστεύω όλοι να φύγουμε από εδώ και να το έχουμε ξεκαθαρίσει, δεν υπάρχει θέμα. Η επικουρικότητα και η αναλογικότητα νομίζω και αυτά είναι θέματα τα οποία ξεκαθαρίζονται σιγά σιγά ότι δεν φύγονται από την οδηγία. Ε, αναφέρθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι συνάδελφοι Α το κρατήσουν στο μυαλό του οι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια για τι συζητήσει που θα γίνουν στη χώρα μέλη του. Και επίση ε, ήθελα να επισημάνω το 40% δεν είναι ο δεσμευτικός στόχος, είναι ένα μήνυμο. Μακάρι οι χώρες να μπορέσουν να εγγυηθούν το 50%. Ε, είναι ένα μήνυμο όμως του διαφορετικού φύλου. Διότι πρέπει να επισημάνουμε, στην έρευνα που έχουμε κάνει υπάρχουν διοικητικά συμβουλία που έχουν πιο πολλές γυναίκες παρά άνδρες. Εκεί θα πρέπει οι άνδρες, στο, το ανδρικό ποσοστό να αυξηθεί. Μίνιμουμ 40% στο κάθε φύλλο. Τώρα ε, το τελευταίο που θέλω να πω και να κλείσω εδώ κυρία Πρόεδρε, καταλαβαίνω την έννοιαση για το χρόνο, η παρέμβαση αυτή η ευρωπαϊκή που έχει σκοπό να ενισχύσει την ε, ενιαία αγορά και τον τρόπο που λειτουργεί και επίσης να δώσει μια όθηση σε χώρες που δεν έχουν ακόμη ασχοληθεί με το θέμα και που διστάζουν ακόμη περισσότερο. Δεν ενοχλεί τις χώρες που πιστεύουν ότι με, τα, με τις μεθόδους που έχουν υιοθετήσει θα τα καταφέρουν. Αυτό κρατήστε το κατά νου, κυρίως οι χώρες που είναι αισιόδοξε για τις μεθόδους τους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, αν είναι τόσο πεπισμένες ότι η αυτορύθμισή τους θα φέρει τα αποτελέσματα αυτά που τα δέχονται ότι είναι νόμιμα και λογικά, ε, δεν θα τις ενοχλήσει καθόλου διότι η οδηγία ακριβώς την υποχρεωτική αυτορύθμιση θέλει να προχωρήσει με συγκεκριμένο στόχο. Ας δώσουν όμως την ευκαιρία σε άλλες χώρες να υιοθετήσουν εργαλεία που θα τις πρόξουν μπροστά αφού από μόνες τους δεν μπορούν να τα καταφέρουν σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ um ε, μου ζητήσατε να είμαι σύντομη, οπότε συμφωνώ απολύτως με την κυρία Κράτσα και θα ήθελα και άρα και εγώ να ευχαριστήσω και εσάς, ε, τους εθνικούς βουλευτές και ε, επί της ουσίας να πω το εξής. Το θέμα εδώ πέρα είναι πραγματικά να ρίξουμε λίγο φως στο σκοτάδι, δηλαδή στο σκοτάδι των διαδικασιών επιλογής, να είναι πιο διαφανής και να μην έχουμε μόνο τις χρυσές φούστες, αλλά να δούμε τι γίνεται μεταξύ τα παντελόνια. Έχουμε αναλύσει από την Ιταλία που δείχνουν πως μέσω τέτοιων ε, διαδικασιών και υποχρεωτικών στόχων η ποιότητα των διοικητικών συμβουλίων αυξήθηκε. Και ε, τα μέλη που επιλέγονται ήταν γυναίκες και άντρες γιατί είναι πιο διαφανή η διαδικασία, Μία μικρή παρατήρηση ε, προ την κυρία Νίμπλερ όσον αφορά την νομική βάση. Δεν, έχουμε, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να συμπεριλάβουμε και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι μόνο τα μη εκτελεστικά. Τώρα, λοιπόν, θα ήθελα να σας προσκαλέσω να συζητήσουμε άτυπα στη συνέχεια σε ε, ένα μικρό γευματάκι που έχουμε προετοιμάσει εδώ πέρα, κάτι σαντουιτσάκι έξω από την Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τα επιχειρήματα που ακούστηκαν, αυτό το μοσαϊκό εδώ πέρα που σχηματίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τέλος ευχαριστώ και τους διερμηνείς που ε, ξεπέρασαν το ωράριό τους. Ευχαριστώ.